chers collègues, bonjour. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Vous êtes aussi au, au sein de la commission. Είστε στην Επιτροπή Μεταφορών και εύχομαι σε όλους και σε όλες καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθανε και οι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήρθαν στη συνεδρίαση. Εδώ έχουμε ένα μήνυμα από τους διερμηνείς. Οι διερμηνείς σας πληροφορούν με τα λύπης ότι συνεχίζεται η εργασιακή διαμάχη με τη δίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις νέες συνθήκες εργασίας που το αντικείμενο που προειδοποίηση για περιακή κινητοποίηση. Η ποιότητα της Γερμανίας για τους ευρωβουλευτές και τους ευρωπαίους πολίτες κινδυνεύει. Δυστυχώς, λόγω της εργασιακής διαμάχη, η διερμηνία θα σταματήσει στις 18.30 όπω προβλέπει το πρόγραμμα συνεδρίασης. Έχουμε παρόντα λοιπόν πολλά μέλη εθνικών κοινοβουλίων. Ανάμεσα στα μέλη έχουμε και μέλη τη ε, συνέλευση τη Σερβία. Έχουμε ένα θέμα που μα απασχολεί όλου σήμερα. Θέλουμε να προωθήσουμε τα δίκτυα των μεταφορών στην Ευρώπη και το μέλλον του συστήματος κινητικότητάς μας. Λοιπόν, εντός της Επιτροπής μας έχουμε ένα σύστημα, θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών, σύγχρονο είναι πρωταρχική σημασία γιατί επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες και στα αγαθά μας να κυκλοφορούν εντάχει με ευκολία μέσω των χωρών της Ενώσεως αλλά και να μπορούμε να συνδεόμεθα και με τους γειτονέ μας και με πιο μακρινές χώρες. Έχουμε και στόχους ε, σε σχέση με το κλίμα, κοινωνικούς στόχους, ενεργειακούς στόχους, πάνω απ' όλα έχουμε στόχο την υπηρεσία, διότι πρέπει να είναι βασικό κλειδί, στοιχείο κλειδί οι μεταφορές για να μετακινούμεθα. Θέλουμε να προετοιμάσουμε να προλιάνουμε το έδαφος για την κινητικότητά μας, μια βιώσιμη κινητικότητα θέλουμε και είμαι πεπισμένη ότι θα τα καταφέρουμε προσανατολιζόμενοι προς καινοτομίε και μέσω αλληλεγγύης να πετύχουμε τους στόχους μας και η πολιτική του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, το RTT, που υιοθετήθηκε το 2013, έχει στόχους, αυτούς που ανέφερα, και πρέπει να έχουμε συντονισμένε προσπάθειε που καταβάλουμε σε όλα τα επίπεδα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο να καταβάλλονται προσπάθειε, καθώ και σε περιφερειακό επίπεδο. Μα μένει ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε με κάθε κατάλληλη προσπάθεια να προσανατολίσουμε σωστά τις επενδύσεις και μέσω των δημοσίων προϋπολογισμών να παράσχουμε την αναγκαία υποστηρίξη στην υλοποίηση αυτών των ε, δικτύων. Λοιπόν, οι επενδύσει που θα διατίθενται για τι ευρωπαϊκέ μεταφορέ, κατά πολύ εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη καθώ και από την υποστηρίξη των προγραμμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι ο μηχανισμό διασύνδεσης ε, τη Ευρώπη. Όμω, ε, όπω γνωρίζετε, ο προπολογισμό τη Ένωση μετά το 2020 επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων και ο προπολογισμό αυτός θα καθορίσει τα μέσα που θα διατεθούν για επενδύσεις σε υποδομές των μεταφορών. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις μέσω δύο συζητήσεων. Θα συναντηθούμε και με τον κύριο Έττιγκερ, που είναι ο επίτροπος επιφορτισμένος με θέματα προπολογισμού και ανθρωπίνων πόρων, ο οποίος θα καταφτάσει και έτσι θα μπορέσουμε να μάθουμε ακριβώς ποιο θα είναι ο προσανατολισμό που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίω στον ε, τομέα των μεταφορών. Πριν ξεκινήσουμε, πριν αρχίσουμε το πρώτο τμήμα συζητήσεων να υποδεχτώ στην Επιτροπή μας μια αντιπροσωπεία από τη Μολδαβία, μια περιοχή που είναι στη Ρουμανία Είστε εκεί, μπορείτε να σηκωθείτε παρακαλώ. Καλώ ήρθατε, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα. Μπορούμε να του χειροκροτήσουμε, του φιλοξενούμενου μα. Και θα ξεκινήσει το πρώτο τμήμα των συζητήσεων που αφορά τα δίκτυα των μεταφορών. Ποια είναι η όλη κατάσταση που επικρατεί, ποιε είναι οι προοπτικέ που μα δημιουργεί το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, έχω τη χαρά να υποδεχθώ του ομιλητέ μα τον κύριο Ζαν Λουί Κάλσον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι υπεύθυνο της Μονάδας για Επενδύσεις, ο κύριος Κόλσον και για τις μεταφορές εντός της Γενικής Διευθύνσεως ΜΟΥΒ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή μας. Τον κύριο Μάτιο Γκρός, ε, είσαστε συντονιστής όσον αφορά το διάδρομο του κεντρικού δικτύου που συνδέει με τη Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη Χαιρόμαστε που μας θυμάστε. Ο κύριος Δανιέλ Ιμπανές, οικονομολόγος και θα εστιαστείτε. Ανακοίσαστε. Θα αναφερθείτε κυρίω στα θέματα αυτά τα οικονομικά. Μας τιμάτε που δείχνει την πρόσκλησή σας και χαίρομαι που είναι εδώ και ο κύριος Μάρκ Βαν Ντάικ, επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων του ε, λιμανιού του Ρότερνταμ σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας και για να οργανώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ε, συζητήσεις θα καλέσω τους συμμετέχοντες των Εθνικών Κοινοβουλίων να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής. Είναι διαφορετικών χρωμάτων αυτά τα έντυπα για τις δύο συνεδριάσεις και για το χρόνο ερωταπαντήσεων παρουσία του Επιτρόπου. Θέλουμε να είναι δυναμική ανταλλαγή των απόψεων και για τους Ευρωβουλευτές όσοι ήθιστε θα αρκεί για σας, όπως κύριε Βιν Βαντεκάμπ να σηκώσετε το χέρι σα. Αυτό αρκεί. Δεν έχετε να συμπληρώσετε έγγραφο. Απλώς σηκώνετε το χέρι. Είναι αρχές απογεύματο, να το ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν για αυτά. Παρακαλώ να είστε λακωνικοί, ούτως ώστε να τροφοδοτηθεί η συζήτηση και όλοι να μπορούν να συνεισφέρουν η παρέμβαση των βουλευτών, σας το λέω ειλικρινά αγαπητοί συνάδελφοι, θα περιοριστεί σε δύο λεπτά. Εγώ ελέγχω το χρόνο, λέω δύο λεπτά είναι δύο λεπτά. Τελειώσατε, τελειώσατε, σας κόβω το μικρόφωνο στα δύο λεπτά. Σας προειδοποίησα. Ακριβώς για να μπορέσουν να μιλήσουν όσων δυνατόν περισσότεροι. Και θα λάβω υπόψη μου και τους αγαπητούς διερμηνείς θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα για να σεβαστούμε το χρόνο στη διάθεσή μας. Και παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων, αν είχα την καλοσύνη να μην μιλάτε πολύ γρήγορα να παίρνετε το λόγο για να μπορούν να σας μεταφράζουν διερμηνείς. Παρακαλώ τους ομιλητές εδώ που είσαστε εδώ να σας πω ότι πρέπει και εσείς να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσης για να υπάρχει περιθώριο για συζήτηση. Και μετά τις παρουσιάσεις θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις των εθνικών βουλευτών, μετά των Ευρωβουλευτών και θα καλέσουμε όλους τους βουλευτές που θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση να το γνωστοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που θέλουν να λάβουν το λόγο κατά τη συζητήσεω θα πρέπει να συμπληρώσουν, το επαναλαμβάνω αυτό, το έντυπο εγγραφή, το γαλάζιο έντυπο και να το δώσουν ε, στους ε, Κλητήρε. Είναι σαφή η κανόνα του παιχνιδιού. Ναι. Όλοι καταλάβατε, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αμέσως λοιπόν από τον πρώτο, τον κύριο Κόλσον. Κύριε Κόλσον, έχετε το λόγο. Επτά λεπτά. Χρονόμετρο, το ξεκινάω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντελή. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας εδώ. Και σας ευχαριστώ που σήμερα συγκεντρώσετε ευρωβουλευτές και εθνικούς βουλευτές. Όντως, η σχέση μεταξύ της εθνικής δράσης και της ευρωπαϊκής δράσης όσον αφορά την πολιτική μεταφορών και υποδομών είναι πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό το ότι βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί είναι κέρια σημασία. 25 χρόνια τώρα υπάρχει η πολιτική αυτή και νομίζω ότι έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές. Πρώτον, η κατάσταση και η πρόσβαση στις υποδομές μεταφορών, οδικές, ε, εσωτερικών υδάτων κτλ. μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που έχει ενισχυθεί κατά πολύ. Δεύτερον, η σύνδεση στα εθνικά σύνορα επίσης έχει προθεθεί πολύ, κάτι το οποίο δημιούργησε άνευ προηγουμένου δυνατότητες για περιφερειακή συνεργασία. Επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω για παράδειγμα Πρατισλάβα Βουδαπέστη ή Κοπεχάγη Μάλμο. Τρίτον, μια ισορροπημένη ανάπτυξη των υποδομών έχει διασφαλιστεί παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις γειτονές χώρες που έχουν συμμετάσχει. Τέταρτον, 10.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων δημιουργήθηκαν, κάτι το οποίο αποτελεί τεράστιο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αν οι πολίτε το θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό πια, όπως επίσης και οι επιχειρηματίε που ταξιδεύουν. Έπειτα, οι υπηρεσίε διαχείρισης τη κυκλοφορία έχουν δημιουργηθεί και για τα εσωτερικά ύδατα και για τις οδικές μεταφορές. Επίσης, η διασύνδεση ανάμεσα των διαφόρων μορφών μεταφορών και για το, τις εμπορικές μεταφορές και για τις επιβατικές είναι κάτι που έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται και σε εθνικό επίπεδο. Τέτοιες εξελίξεις βέβαια εξαρτώνται από την δέσμευση που παίρνουν πρώτα απ' όλα οι χώρες μέλη. Γιατί πράγματι οι υποδομές μεταφορών αποτελούν σημαντική επένδυση για κάθε χώρα μέλος και η υλοποίησή τους εξαρτάται από τους εθνικούς κανόνες και τις διαδικασίες. Πάντω, η πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων σίγουρα προσφέρει μια επιπλέον ευρωπαϊκή προοπτική, επιπλέον από την εθνική, με αποτέλεσμα ωφέλη για ολόκληρη την Ευρώπη. Οφέλη, το οποίο είναι μεγαλύτερα από ότι αν συσσωρεύαμε με μονομένες δράσεις εθνικού επίπεδου. Η σημερινή πολιτική που ξεκίνησε το 2013 για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ξεχωρίζει τα διάφορα δίκτυα προκειμένου να επικεντρωθεί σε δίκτυα τα οποία έχουν μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για να πετύχουμε το στόχο της συνοχής, της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και οφελών για όλους τους πολίτες. Θέλουμε δηλαδή να γενικεύσουμε το πλαίσιο το επενδυτικό σε εποχές δύσκολες δημοσιονομικά. Μετά από έξι χρόνια λοιπόν εφαρμογή τη νέα πολιτική διευρωπαϊκών δικτύων, νομίζω ότι πλέον να αντιμετωπίσουμε τι εξή προκλήσει. Χρηματοδότηση. Η νέα πρόταση για την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη με τον προπολογισμό που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο προσπαθούν ακριβώς να πετύχουν βελτίωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, μια που είναι το θέμα του δεύτερου πάνελ σήμερα. Έπειτα, συνεργασία, διασυνοριακά και με συμμετοχή πολλών και διαφορετικών φορέων και σε περιφερειακό και σε τοπικό μάλιστα επίπεδο. Αυτό είναι και το κύριο καθήκον των Ευρωπαίων συντονιστών ο κύριος Γκρός και ο κύριος Σίμψον είναι από αυτούς και θα σας μιλήσουν σήμερα για το δικό τους έργο. Τρίτη πρόκληση, τρίτη δυσκολία που έχουμε μπροστά μας είναι πώς θα προωθήσουμε μεγαλύτερα αλλά και μικρότερα προγράμματα. Οι Ευρωπαίοι συντονιστές έχουν δείξει ότι υπάρχει μια συνδυασμένη προσέγγιση και αυτό φάνηκε στην τελευταία κρόση της Επιτροπής Τραν το Φεβρουάριο που μας πέρασε. Τέλος, συμμόρφωση των διευρωπαϊκών δικτύων για να συνδυαστούν με τις άλλες πολιτικές, την διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια, την βιωσιμότητα και την προστασία. Για παράδειγμα, πόσο θα ενισχύσουμε τις υποδομές έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν εναλλακτικά καύσιμα. Και έτσι κι αλλιώς κάτι τέτοιο θα μπορεί να έχει αξία μόνο εφόσον υπάρχει συνέχεια, γιατί το βρίσκουμε σε όλες τις χώρες μέλη, διασυνοριακά. Έπειτα, στο επόμενο ΣΕΦ, την επόμενη διευκόλυνση δηλαδή, ακριβώς πρέπει να προσέξουμε αυτό το θέμα των υποδομών και πώς θα διασφαλίζονται διασυνοριακά. Εδώ πάλι είναι οι Ευρωπαίοι συντονιστέ που έχουν να παίξουν ρόλο, γιατί μπορούν να δώσουν όθηση σε πρωτοβουλίε προς αυτή την κατεύθυνση. Αγαπητοί αξιότιμοι ευρωβουλευτές, η πολιτική των ευρωπαϊκών δικτύων που συνδυάζει παρεμβάσει τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε εθνικό επίπεδο, συντονισμένα, είναι το καλύτερο παράδειγμα πολιτικής που έχει να παρουσιάσει σημαντικά επιτεύγματα. Και επιτεύγματα μάλιστα απτά και γι' αυτό ορατά τα διαπιστώνουν, τα βλέπουν οι πολίτες μας. Οπότε, έχω εμπιστοσύνη ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να στηρίξετε την πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη και θα μας βοηθήσετε και στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόλσον. Συνεχίζουμε. Εσείς κύριε Γκρός, για 7 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Για να σας εξηγήσω ποιος είναι ο ρόλος των συντονιστών, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο για τους εννέα διαδρόμους που έχουμε στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Έχουμε νέα συντονιστές και άλλους δύο, ο Μπραν Σίμψον για παράδειγμα είναι εδώ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις οριζόντιες υποθέσεις, δηλαδή τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας όπως τους λέμε και το ETMS, που αποτελεί βέβαια μια τεράστια πρόκληση. Όπως καταλαβαίνετε είμαστε εδώ ώστε στα πλαίσια του 2030 να έχουμε πετύχει αυτούς τους ε, ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους όπως τους λέμε, να πετύχουμε ανάπτυξη, να πετύχουμε απασχόληση, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί οι μεταφορές πρέπει να κάνουν σημαντικές προσπάθειες. Τώρα για το δικό μου τον διάδρομο, εγώ είμαι υπεύθυνο για το Orient East Med, που ξεκινάει από τη Βόρεια Γερμανία και περνάει από 8 χώρες και φτάνει στην ε, Ελλάδα και προστίθεται και η Κύπρος. Στην τελευταία περίοδο, 80% των επενδύσεων πήγανε στους σιδηροδρόμους. Περιμένουμε οι επενδύσεις αυτές να καρποφορήσουν, ε, εννοείται, ώστε να περάσει η κυκλοφορία από τις οδικές μεταφορές του σιδηροδρόμους. Όλα αυτά τα χρήματα ε, διατέθηκαν από τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Περιμένουμε να υπάρξει η χρήση των κονδυλίων κατά 90%. Οπότε, εδώ δεν είναι για να πούμε ότι χρησιμοποιούμε όλα τα χρήματα, αλλά είναι για να πούμε ότι χρησιμοποιήθηκαν με σωστή οργάνωση έχουμε έτοιμα 410 προγράμματα και τα μισά έχουν ήδη οριμάσει και μπορούν να υλοποιηθούν στην επόμενη περίοδο. Αυτό είναι το έργο μας ως συντονιστές, να συνδέουμε την Ευρώπη, να συνδέουμε δηλαδή τους ανθρώπους και να προετοιμάσουμε μια Ευρώπη ώστε να συνδέεται και με τον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό τα λιμάνια ε, στη θάλασσα, τα αεροδρόμια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα υπάρξουν και τέτοιες χώρες στο μέλλον. Οπότε θέλουμε να υπάρχει συνοχή στα δίκτυα τα οποία προετοιμάζουμε. Η διακυβέρνησή μας τώρα είναι πολυεπίπεδη. Εννοείται ότι ο κύριος συνομιλητή μας είναι οι χώρε μέλη. όμως έχουμε και συνομιλητέ σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο τοπικό. Και γι' αυτό ακριβώ και επιμένουμε ότι η αποδοχή ενός προγράμματος εξαρτάται και από τις πληροφορίες που μαζί δίνουμε εμείς με τις χώρες, με τις περιφέρειες για κάθε πρόγραμμα και για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι σχετικές επενδύσεις. Θα λέγω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλος αυτός του συντονιστή να μην είναι κάτι που βλέπουμε όπως είχε πει κάποιος συνάδελφος ότι δεν είμαστε δικτάτορες, είμαστε για να διευκολύνουμε τα πράγματα. Δημιουργούμε λοιπόν κινητοποίηση γύρω από ένα πρόγραμμα, δημιουργούμε συνεργασία δημιουργικότητα και με συγκεκριμένες εμπειρίες που διαθέτουμε δίνουμε και συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων. Για κάθε διάδρομο, τέσσερις φορές το χρόνο, οργανώνουμε αυτό που λέμε φόρουμ, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι διαφορομενοί φορείς. Είναι μια ανταλλαγή που γίνεται μεταξύ των διαφόρων φορέων και μαζί προετοιμάζουμε το work plan, όπως το λέμε. Εδώ, κυρία Πρόεδρε, μπορώ ήδη να σας δώσω το τελευταίο τεύχος. Έχουμε το τρίτο για τον κόριντορ, τον δικό μου, που περιλαμβάνει προτάσεις για την επόμενη περίοδο. Όταν λοιπόν μιλάμε για οικονομικά στοιχεία, του ΣΕΦ κλπ, δεν μιλάμε μόνο για χρήματα, μιλάμε για συγκεκριμένα προγράμματα επίσης που υπάρχουν στο σχέδιο αυτό που σας έδωσα. Και σε καθένα από αυτά, να ξέρετε, πρέπει να υπάρχει υπογραφή από κάθε Υπουργό Μεταφορών κάθε χώρας. Άρα δεν είναι μια δικτατορία, δεν είναι ένα διάταγμα που έρχεται από πάνω για να εφαρμοστεί, ούτε πρόκειται για ένα μπέρδεμα προγραμμάτων. Είναι σε συντονισμό με τις χώρες μέλη. Και τελευταία παρατήρηση είναι ότι η διαλειτουργικότητα είναι πολύ σημαντικό κριτήριο για την Ευρώπη. Στου σιδηροδρόμους είναι που έχουμε τα περισσότερα προβλήματα. Δίνουμε όμως πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο να έχουμε τεχνικά πρότυπα ευρωπαϊκά μεσοπρόθεσμα. Αυτό θα αποτελέσει και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών και της κινητικότητας στην Ευρώπη. Και αυτό ακριβώς είναι που θα βοηθήσει την Ευρώπη να βρει τη θέση της στην έρευνα παγκοσμίω. Άρα λοιπόν είναι διπλό το όφελος. Πέρα από τα τεχνικά κριτήρια, στο οποίο δίνουμε μεγάλη σημασία. Το RTMS, για παράδειγμα, το σύστημα ε, σημάτων, σηματοδότησης. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία όχι μόνο στις επενδύσεις, αλλά στην αποτελεσματικότητα των μεταφορών που εξαρτάται από κανόνες λειτουργίας. Και το παράδειγμα που δίνω στο δικό μου διάδρομο είναι ότι όταν πάρετε στο Αμβούργο το τρένο για να κατέβετε και να πάτε στην Ελλάδα, έχετε 20 ώρες αναμονή στα σύνορα κατά μέσο όρο. Η επένδυση ενός δισεκατομμυρίου παραπάνω για να κερδίσουμε μία ώρα είναι αυτό που μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε σε κάθε πέρασμα συνόρων, να φτιάξουμε μια ομάδα εργασίας που να κοιτάξει τι συμβαίνει και να δώσει συγκεκριμένα, συγκεκριμένες ιδέες, ώστε 20 ώρες να γίνουν δύο. Οι μεταφορές λοιπόν εδώ σε πολλές διαφορετικές περιοχές, τόσο κοινωνικά όσο οικονομικά και πολιτικά, μπορούν να δείξουν ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας στην Ευρώπη. Εμείς αυτό το βλέπουμε στον δικό μας διάδρομο και το βλέπουμε επίσης και όταν εξηγούμε τα ωφέλη της κοινή προσέγγισης. Οι διασυνοριακές μεταφορές είναι το κατεξοχήν παράδειγμα όπου η Ευρώπη πρέπει να παρέμβει έχουμε κέρδος. Η προστιθέμενη αξία είναι το ότι επενδύοντας στην Ελλάδα ή στη Ρουμανία είναι κάτι από το οποίο μπορεί να υποφεληθεί τον Βούργο ή ξέρω εγώ ποια άλλη περιοχή της Ευρώπης. Και σε αυτό επιμένουμε και υποστηρίζουμε ακριβώς αυτή την προσέγγιση. Ελπίζω στο μέλλον και οικονομικά, αλλά και όσον αφορά τις επαφές με διάφορες χώρες μέλη, να είμαστε εξίσου καρποφόροι. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρό. Ο κύριος Λιμπανέ, ο επόμενο ομιλητή μα έχετε και διαφάνειε. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας πρώτα, έτσι. Έχουν αρχίσει να προβάλλουν διαφάνειες. Ωραία. Ευχαριστώ. Παρόλο που αυτό το πρόγραμμα είναι από τα ακριβότερα στην Ευρώπη, ε, δεν είναι και τόσο γνωστά από τους πολίτες Ευρώπης. 26 δι. Οπότε το θέμα είναι τι γίνεται τώρα με τις δεσμεύσεις τη ε, οικονομικές της Γαλλίας και της Ιταλίας. Τη στιγμή που προ το παρόν έχουμε μόνο να δεις ε, επενδύσεων για να τεκμηριωθεί αυτό το πρόγραμμα, αυτό το έργο. Αλλά δεν προχωράνε διαφάνειες όμως. Πήγαμε στην επόμενη, τέλο πάντων. Για να τεκμηριωθεί λοιπόν αυτό το έργο έχουν προβλεφθεί αύξηση των ροών των επιβατών και των εμπορευμάτων. Για το 1991 είχαμε υψηλότερε προβλέψει από την πραγματικότητα. Για το 2000 για το 2000 αντίστοιχα 40% λιγότερε προβλέψει. Βάσει λοιπόν αυτών των προβλέψεων το έργο αυτό ξεκίνησε το 2006 είχαμε νέες προβλέψεις, ακόμα πιο μακριά την πραγματικότητα. Για το 2017 θα είχαμε πάνω από 3 εκατομμύρια βαρέα οχήματα και πολλά εκατομμύρια εμπορευμάτων. Για το 2017 λοιπόν η πρόβλεψη ήταν 61 εκατομμύρια τόνων ε, εμπορευμάτων, τη στιγμή που είχαμε μόνο 22, δηλαδή το 1 τρίτο της πρόβλεψης. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία η Γάλλο Ιταλική έδειξε πριν από την κρίση ότι το εμπόριο εμπορευμάτων είχε υποχωρήσει. Μιλάμε για την. Α μιλήσουμε τώρα μάλλον για την Ελβετία και την Αυστρία. Εδώ δείχνει το γράφημα ότι οι συνθήκε εδώ είναι τελείω διαφορετικέ. Για πολλά χρόνια οι Ελβετία και οι Αυστριακή απέδειξαν ότι μπορούσαν να μεταφέρουν εμπορεύμα, εμπορεύματα και να εκμεταλλευτούν την υπάρχουσα διαδρομική δομή. Η Γαλλία με τι ίδιε υποδομέ δεν έκανε δεν σημαίνει παρά υποχωρήσεις ε, και στα όρη αλλά και ε, στα παιδινά. Οι μεταφορές βορρά-νότου αυξήθηκαν μέσω της Ελβετίας επειδή είχαμε αύξηση του ΑΕΠ και οι γαλλοϊταλικές μεταφορές μειώθηκαν επειδή ακριβώς μειώθηκε και η βιομηχανική παραγωγή λόγω της μετανάστευσης των βιομηχανιών. Το 92 λοιπόν ξεκίνησε αυτό το έργο και θα μπορούσε να ωφελήσει παρά μόνο σε περίπτωση όπου η Γαλλία και η Ιταλία είναι σε θέση να κάνουν τα ίδια που έκαναν οι Ελβετοί και οι Αυστριακοί με τους ιδεοδρόμους τους. Όλα αυτά είναι πολύ γνωστά και αποδεκτά από τους ίδιους τους ε, σχεδιαστές του έργου. Έχουμε τούνελ τα οποία δεν ε, είχαν λόγο ύπαρξης. Ε, έχουμε τούνελ τα οποία δεν ήταν κατάλληλα κλπ. κλπ. Ο κ. Φεγέτα, ε, εκ μέρου τη Ιταλική κυβέρνηση, είπε το 2017 ότι είναι ένα αφισβήτητο ότι όλε οι προβλέψει που είχαν γίνει, τρέχει πάρα πολύ ο μιλητή, δυστυχώ λυπούμαστε, όλε οι προβλέψει λοιπόν είχαν de facto διαψευστεί. Για τη Γαλλία και την Ιταλία έγιναν απίστευτα πράγματα για να προωθήσουμε το εμπόριο, ε, το ε, εμπόριο εμπορευμάτων, αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Έχουμε υψηλά διόδια στα τούνελ και οι μεταφορείς είδαν ότι είχαν κόστος 30% υψηλότερο στον άξονα αυτό Γαλλίας-Ιταλίας η υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή που από το 80 περιλαμβάνει 37 τρένα πορεμάτων και 40 τρένα επιβατών. Ήταν απλή γραμμή και έγινε διπλής κατεύθυνση. Είχαμε ατμομηχανές που έχαναν μια μισή ώρα και με το νέο υλικό βέβαια από το 2003 δεν χρειάζεται να αλλάζουν. Έχουμε έλεγχο στα τελωνία ε, όπου δεν υπάρχουν πια και κερδίσουμε άλλες ε, δύο ώρες. Τα τούνελ ε, μεγαλήθηκαν, ε, μεγα, μεγάλωσαν και παρόλα αυτά έχουμε έξι φορές λιγότερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. Έχουμε τη μεταφορά ενός εκατομμυρίου φορτηγών μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας στο σιδηρόδρομο. Υπό αυτές λοιπόν συνθήκες, η δυνατότητα των υπαρχουσών υποδομών δείχνει τα εξής. Έχουμε και πάλι ξαναλέω πάνω από ένα εκατομμύριο φορτηγά τα οποία θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε από τους δρόμους ενισχύοντας την υπάρχουσα υποδομή δωρεάν. Θα μπορούσαν δηλαδή από τώρα η Γαλλία και η Ιταλία να πετύχουν τον στόχο του 2050 της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το 50% κυκλοφορία μέσω σιδηροδρόμων. Κανείς δεν αφισβητεί. Κανεί δεν αμφισβητεί λοιπόν ότι έχει επιβληθεί στην, κάτι στην Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Έχουμε στι συνθήκε ε, γύρω στα 50 άρθρα. Έχουμε και ένα μόνο για τη χρηματοδότηση. Έχουμε μια ανταλλαγή μεταξύ Γαλλία και Ιταλία. Και στι συνθήκε δεν υπάρχει ουδέμια ρήτρα παράβαση. Υπάρχουν μόνο κάποιες ενδείξεις και οι μόνες ενδείξεις αφορούν ακριβώς την, ε, τις υπάρχουσες ε, ε, συνδρομικές διαδρομές. Πρέπει λοιπόν το, το θέμα αυτό να το δούμε στο σύνολό του. Η δεσμεύση της Γαλλίας και της Ιταλίας είναι να οικοδομήσουν το κοινό τμήμα το οποίο όμως αφορά το διασυναριακό τούνελ. Η Γαλλία δεσμεύτηκε να χτίσει με δικά της έξοδα 14 χιλιόμετρα τούνελ παραπάνω από την Ιταλία αν η Γαλλία λοιπόν δεν χτίσει αυτά τα 33 χιλιόμετρα που πρέπει, τότε η Ιταλία μπορεί να αρνηθεί να πληρώσει το δικό της μερίδιο. Πρέπει τα χιλιόμετρα αυτά με τούνελ να είναι διαθέσιμα πριν από την έναξη των τελικών εργασιών και μάλιστα το κόστος των έργων θα πρέπει να πιστοποιηθούν από τρίτους και αυτό είναι το πρωτόγνωρο. Όπως βλέπετε οι συνθήκες δεν τηρούνται. Τίθενται κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν κάποιες πρακτικές σε αυτό τον φάκελο και θα δείτε εδώ κάποια παραδείγματα είναι εδώ στην ε, είσοδο της αίθουσα. Αυτά βεβαίως αφορούν τους ε, εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους βουλευτές και τους υπόλοιπους υπαλλήλου. Αυτές οι εργασίες λοιπόν παρουσιάστηκαν ως προκατακτικά έργα για να λάβουν 50% ε, προκαταβολών αντί 40% τη στιγμή που το έργο δεν ήταν έτοιμο. Μπορούμε λοιπόν να να ζητήσουμε να εξεταστεί αυτό το χρέος. Αλλά τι γίνεται με τις προβλέψεις για το υπόλοιπο χρέος, το οποίο είναι μη εφικτό, ανέφικτο. Είχαν 58% επιδοτήσεις, 28 εκατομμύρια ευρώ κόστος ανά χιλιόμετρο. Οπότε ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την ε, για αυτόν τον εκτροχιασμό τον δημοσιονομικών των δύο χωρών. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όλες οι γαλλικές διοικήσεις απέρριψαν τη την ε, σύνδεση με το Τωρίνο και κηρύχθηκαν σε οικονομικά μειονεκτική θέση. Θα πρέπει λοιπόν να τηρηθούν οι, οι συνθήκες για τη σύνδεση με το Τωρίνο στο μέλλον. Θα πρέπει να εργαστούμε ώστε να μειώσουμε την κυκλοφορία ε, εμπορευμάτων, κάτι το οποίο ήδη είναι εφικτό από σήμερα. Και σας καλώ να κοιτάξετε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχω επισυνάψει στο φάκελο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ την Επιτροπή και ευχαριστώ τους καημένους ερμή οι οποίοι υπέφεραν με την παρουσίασή μου. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Βανδίκ, επικεφαλής των εξωτερικών σχέσεων, εξωτερικών υποθέσεων του λιμανιού του Ρότερνταμ. Έχετε το λόγο. Και εγώ έχω κάποιες διαφάνειες. Ίσως να πάρω το τηλεχειριστήριο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους που με καλέσατε. Μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Να μιλήσω λίγο για το λιμάνι του Ρότερνταμ και το ρόλο των λιμανιών στους διαδρόμους. Το λιμάνι του Ρότερνταμ λοιπόν είναι μεγάλο λιμάνι στα βορειοδυτικά της Ευρώπης, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε ποτέ το μεγαλύτερο λιμάνι αν ασχολιόμασταν μόνο με την Ολλανδική αγορά. Χρειαζόμασταν την Ευρωπαϊκή αγορά και η εσωτερική αγορά μας διευκόλυνε για να επεκταθεί το λιμάνι του Ρότερνταμ στο βαθμό που μεγάλωσε. Θα πρέπει να καταλάβουμε βλέποντας τους αριθμούς ότι έχουμε σημαντικό ρόλο στην περιοχή για την απασχολησιμότητα, για το εργατικό δυναμικό. 180.000 άνθρωποι άμεσα και έμεσα εργάζονται για το λιμάνι και για την ευρύτερη περιοχή και έχουμε και μεγάλη συνεισφορά όσον αφορά το ΕΠ της Ολλανδίας. Βλέπετε μια εικόνα εμπορευματοκιβώτια, μακροοικονομική πολιτική είναι πολύ καλά, τα κιβώτια αυτά είναι 30% ε, των νεκρών από το λιμάνι, αλλά έχουμε ακόμα τα μεγάλα αγαθά Έχουμε 9 εγκαταστάσεις, 5 ε, δηληστήρια και 30 χημικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι. Έχουμε λοιπόν, ε, είμαστε κόμβος βιομηχανικός και επιμελητίας. Ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων λείπει εδώ. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολλά που κινούνται μέσα στο λιμάνι. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα λιμάνια. Αν μιλήσουμε για το Αμβούργο, την Αμβέρσα, Μασαλία, και Βαλένσια. Είναι κόμβοι, βιομηχανικά λιμάνια, οργανωτικά. Βλέπετε την κάλυψη των διαφόρων περιοχών. Το πορτοκαλί είναι Χαύρι και Αμβούργο, Αμβέρσα και Ρότερνταμ. Δεν καλύπτουν μόνο τις χώρες τους αυτά τα λιμάνια, αλλά όλη την βορειοδυτική Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για τα βαλτικά λιμάνια, τα λιμάνια της Αδριατικής, που καλύπτουν τη δική τους περιοχή. Βλέπετε σημαντικό διασυνοριακό ρόλο που έχουν τα λιμάνια στον φορά των εμπόριο και έχουν και επιρροή διασυνοριακή. Το Ρότερνταμ συνδέεται με τρεις διαδρόμους, Ρίν, Άλπη, Βόρεια Θάλασσα, Μεσόγειο, Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική. Είναι κρίσιμο θέμα για μας και είναι σημαντικό μήνυμα από εμά. Συνεχίστε την ε, πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων, όπως έγινε και τώρα, πολύ ορθολογική πολιτική που ξεκίνησε το 2013 για την αύξηση ανταγωνιστικότητας τη Ευρωπαϊκή αγοράς, ε, δημιουργώντα τι κατάλληλε υποδομές, βασικές υποδομές. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και προκλήσεις. Αν δείτε λοιπόν ε, πώς 48% γίνεται με φορτηγά η μεταφορά στο λιμάνι, 42% των μεταφορών γίνονται ε, με μαούνες και εσωτερική ναυσοπλοεία και 12% με σιδηροδρόμους μεταφέρονται τα εμπορεύματα και πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό των σιδηροδρόμων τα επόμενα χρόνια όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρόκληση. Βλέπετε τι είδου προγράμματα προωθούμε. Βλέπετε μια γέφυρα στην εικόνα, δείτε καλά, δεν υπάρχει ακόμα, κατασκευάζεται. Είναι από τα βασικά μας προγράμματα που σηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω διευρωπαϊκών δικτύων ε, και ε, θέλουμε να περνάνε τα εμπορεύματα από τον ΜΑΣ στην ανοιχτή θάλασσα και τα προϊόντα που έρχονται από τη Γερμανία να πάνε στο λιμάνι. Στη Γερμανία υπάρχει το πρόβλημα επίσης ε, να υπάρξει σωστή διασύνδεση, αλλά αυτό είναι θέμα χρόνου. Όσον βλέπετε το κομμάτι του ThemesVec, προσπαθούμε να, τον, να, έχουμε μεταφορές μεταξύ Ρότερνταμ και ενδοχώρας για να τονίσουμε ε, τους διάφορους, διάφορους κόμβους μεταφορών, επενδύει το λιμάνι του Ρότερνταμ στις διασυνδέσεις για να στηρίξει τους εμπορευόμενους, για να υπάρξει μεταφορά εμπορευμάτων, διασύνδεση με, άλλα, με άλλες περιοχές. Λοιπόν, μετακίνηση ε, διατροπική και θέλουμε και ψηφιοποίηση για να είναι πιο βιώσιμες οι διασυνδέσεις. Δύο πολιτικές ακολουθούμε. Η μία είναι η ψηφιοποίηση. Οι διασυνδέσεις με τον ενδοχώρα πρέπει να βελτιστοποιηθούν. Πρέπει να κινούνται οι πληροφορίες μεταξύ των εμπλεκομένων προηγουμένων. Φαίνονται λογικά αυτά αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να λυθούν όλα αυτά και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λογική αυτοματοποίηση των μεταφορών. Είναι προτεραιότητα για τα επόμενα έτη. Θέλουμε να τονώσουμε και εναλλακτικά καύσιμα σε συνεργασία με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το Rotterdam έχει το μεγαλύτερο τερματικό γεγροποιημένο φυσικό αέριο LNG και θα χρησιμοποιηθεί και για ακτοπλοεία και για διαπόντιες διασυνδέσεις ευρύτερα το LNG. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λιμένων, η ΕΣΠΟ, έκανε έρευνα. Πριν από δύο μήνες ξεκίνησε. Νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές έχουν αυτή την εικόνα, οι άλλοι σας όχι θα το στείλουμε ψηφιακά. Επενδύσεις, υποδομές επενδύσει που χρειάζονται και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Ζητήσαμε του χειριστέ, διαχειριστέ των λιμανιών. Τι προβλήματα έχετε για το μέλλον, για τι επόμενε περιόδου. 37% τεράστια προβλήματα δήλωσαν ότι έχουν όσον αφορά επενδύσεις σε βασικές υποδομές. Χρειάζεται να καλυφθούν τα κενά των διευρωπαϊκών δικτύων όσον αφορά και τους διαδρόμους. Και νέες επενδύσεις χρειάζονται για τα ψηφιακά, στον Βούργο Φερρυπίν, επενδύουν και στα δίκτυα 5G και στο Rotterdam επενδύουμε και σε ενεργειακές υποδομές. Ατμό ε, και ε, γεωθερμικές πηγές να χρησιμοποιηθούν, ε, κυρίως η θέρμανση πόλεων. Τέτοιου είδους επενδύσεις ε, και προκλήσεις μας περιμένουν και, και, χρειάζεται και ο διάδρομος διασυντησιμότητας 2.0 να ενταχθεί στα, στα πλαίσια του διευρωπαϊκού δικτύου, των ευρωπαϊκών δικτύων και να κινηθούν προς το μέλλον εστιαζόμενοι επιστηφιακών υποδομών και ενεργειακών που απαιτούνται για μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Βλέπουμε εδώ το διαχωρισμό. Είπα ότι έχουν κρίσιμο ρόλο διασυνοριακό τα λιμάνια με προστιθέμενη αξία κατά το μήκος των διαδρόμων Ξεκινούν και λήγουν οι διάδρομοι με βασικούς κόμβους στα λιμάνια. Στο προηγούμενο TNT μόνο 4% των πόρων πήγαν στα λιμάνια. Το μεγαλύτερο ποσό πήγε στη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμων, το υποστηρίζουμε, πρέπει να γίνει αυτό, αλλά θεωρούμε ότι δεν πήραν αρκετά χρήματα τα λιμάνια. Δεν έχουν αναγνωριστεί ότι βοηθούν και τα λιμάνια καλύτερα τη διασύνδεση με την ενδοχώρα και αυτή είναι η έκκλησή μας την επόμενη ε, περίοδο. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, αν επιτρέπετε σε ένα λεπτό να πω κάποια πράγματα. Βασικά μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε για τις νέες προτάσεις για το νέο μέσο για διασύνδεση της, Ευρω... Ε, της Ευρώπης, το ΣΕΦ2. Μελλοντικές προκλήσεις για τα λιμάνια πρέπει να σημειωθούν και για οργανωτικούς λόγους και επιμελητίας. Χρειάζεται ψηφιοποίηση και αλλαγή όσον αφορά τις ενεργικές πηγές για σύνδεση με την ε, ενδοχώρα. Χρειαζόμαστε πόρους από το ΣΕΦ2 γι' αυτό. Μπορούμε να κάνουμε πολλές έρευνες, αλλεπάλληλες, αλλά βέβαια χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα υλοποίηση. Η υλοποίηση δεν είναι καλά ισορροπημένη. Αν βλέπετε τον ορίζοντα 2020 και το νέο ορίζοντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι 100 προς 42 αναλογία. Χρειάζεται μεγαλύτερη ισορροπία. Τελικό μήνυμα που σας απευθύνω. Αυτονόητο. Χρειάζεται υποδομ... Ε, υποδομές λιμενικές, να επενδύσουμε σε λιμενικές υποδομές και το 40% του προπολογισμού για πιο σύγχρονες επενδύσεις υποδομές σχετικά με ψηφιοποίηση και την αλλαγή της χρήσης των ενεργειακών πηγών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε για το λιμάνι του Ρότερνταμ. Συζήτηση τώρα. Πρώτα απ' όλα, για δύο λεπτά, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπόντα από τη Ρουμανία. Πού είναι? Για να σας δω. Εκεί. Καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πω ευθύς εξ αρχής ότι η Ρουμανία έχει νομοθετήσει όσον αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό για μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών. εντοπίστηκαν ε, διάφορα θέματα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα μεγάλων υποδομών για την περίοδο 2014-2020. Οι επενδύσεις για τις βασικές υποδομές αποτελούν προτεραιότητα για την Ρουμανία στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έχουμε για το ΣΕΦΠΕ μετά το 2020. Πιστεύουμε ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί ένα από τα μέσα χρηματοδότησης από τα πιο σημαντικά για τόσα έχουν γίνει στον τομέα του, των μεταφορών. Εγκρίθηκε ένα κείμενο για τους διαδρόμους μεταφορών που δείχνει ότι το κύριο δίκτυο που προτείνει η Ρουμανία για το 2030 πρέπει όντως να υλοποιηθεί. Ακόμα και αν βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις ανάγκες χρηματοδότησης και τα κονδύλια, τα οποία κατ' έχουν ε, αποφασιστεί για την Ρουμανία. Μιλάω πάντα, όπως σας είπα, για τις βασικές υποδομές. Είμαστε τώρα στα μέσα του δρόμου της περίοδου 2014-2020 ε, το ποσοστό χρήσης των κονδυλίων δεν είναι το επιθυμητό, κυρίως όσον αφορά την απορρόφηση για τον ε, μηχανισμό διάβαση στην Ευρώπη. Όπως ίσως το γνωρίζετε, ο βαθμός ε, απορρόφησης στη Ρουμανία εξαιτίας της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις ήταν κάτι δύσκολο, αλλά η τελευταία κυβέρνηση αποφάσισε να υπάρχει και μια διαδικασία κατεπήγοντος που απλοποιεί τις δημόσιες συμβάσεις, ε, σεβόμενοι όμως βέβαια τα όσα έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 για τις δημόσιες αυτές συμβάσεις. Για την περίοδο πάντα 2014-2020, για πρώτη φορά περάσαμε από διαφορετικά προγράμματα ε, που όπως είχαμε πριν για την Ανατολική Ευρώπη και για τη Δυτική Ευρώπη, σε κάτι νέο για ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό είναι μεγάλη ελπίδα για μένα για μετά το 2020 τώρα, ελπίζω να μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε περισσότερο το θέμα των μεταφορών στην Ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπότ. Πάνω από δύο λεπτά όμως, ε. Προσπαθήστε να τηρείτε το χρόνο σας. Δύο λεπτά ο καθένας. Για να ακούσουμε και περισσότερους. Ο κύριος Πούκης, Λετωνία. Πού είσαστε? Καλώς ήρθατε κι εσείς. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ε, είμαι βουλευτής στο Κοινοβούλιο της ε, Λετωνίας, στην Επιτροπή Οικονομίας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι για την Λετωνία και τις γείτονες χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τις υποδομές μεταφορών. Για τις βαλτικές χώρες, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υλοποιηθεί η διαδρομή της Βαλτικής που θα οδηγήσει στη σύνδεση της Πορτογαλίας με όλη τη Δυτική Ευρώπη. Και είναι και στρατηγική σημασία, αλλά και πολιτικά και οικολογικά και οικονομικά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Προσβλέπουμε λοιπόν στη διαδρομή αυτή και ελπίζουμε να υλοποιηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Θέλω τώρα εσά, κύριε Αντελή, αλλά και του συναδέλφου ευρωβουλευτές στην Επιτροπή σας να ρωτήσω. Πιστεύετε κι εσείς ότι ο σιδηρόδρομος της Βαλτικής είναι όντως ένα από τα προγράμματα που πρέπει να υλοποιηθεί βάσει του προγραμματισμού και να μην υπάρξουν δυσκολίες και να υπάρξει και κατάλληλη χρηματική πρικοδότηση. σε ευχαριστούμε. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνεται να παρακολουθήσουμε τις παρουσιάσεις αυτές που είναι ένα κλασικό παράδειγμα του τι έχει γίνει και τι μας μένει ακόμα να κάνουμε. Είμαι σκιώδη συζητήτρια της ομάδας μου για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο από το 2021. Θέλω λοιπόν να πω ότι όλοι συμφωνήσαμε και εγκρίθηκε για το σχετικό κείμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ότι τα σημερινά ποσά στον προπολογισμό σε σχέση με τις φιλοδοξίες που εντοπίσαμε στο παρελθόν, δηλαδή να υλοποιήσουμε όλους τους διαδρόμους των βασικών υποδομών, και υπάρχουν βέβαια και υπόλοιποι, όλα τα σχέδια, που είναι εξαιρετικά σχέδια τις περισσότερες φορές, το είπε η Επιτροπή, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για τη φιλοδοξία που έχουμε. Τώρα θα το συζητήσουμε και μετά, αλλά θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο σε κάποια ζητήματα. Πια, πραγματικά χρειαζόμαστε τους μεγάλους ε, διαδρόμους και πρέπει να προχωρήσουν με προβολή, με συνένεση και γι' αυτό είναι αναγκαίο να ακολουθήσουμε κανόνες του τρίτου πακέτου κινητικότητας που προσπαθούν να καλύψουν τα ε, διασυνοριακά ζητήματα. Είτε είναι αυτά κανονιστικά, είτε είναι περιβαλλοντικά, είτε έχουν να κάνουν με την διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών κτλ. Δεύτερον, θα έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα, η χρηματοδότηση, να μπορέσει να προσφέρει ευκαιρίες να υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν επιδοτήσεις, άλλοι θέλουν το επενδυτικό μείγμα, το blending, άλλοι θέλουν περισσότερο ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα πρέπει η συγχρηματοδότηση να μην επιβαρύνει ξαφνικά και υπερβολικά το χρέος των χωρών μελών. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε ότι μερικές φορές ο εθνικός προγραμματισμός με τον ευρωπαϊκό να αποτελούν ένα σύνολο. Δεν είναι δυνατό στις Βρυξέλλες να εγκρίνουμε έναν προγραμματισμό, για παράδειγμα αυτό για το τορίνο και μετά για το Παρίσι να μην είναι αυτό προτεραιότητα. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη να θυμίζει στις χώρες μέλη ότι θα πρέπει οι αποφάσεις να είναι ενιαίες στην Ευρώπη και στις χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ορτασούν. Πού είναι? Α, εσείς εκεί, όχι, από τη Σουηδία. Ορτασούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας μεταβιβάσω την δέσμευση της χώρας μου, της Σουηδίας, για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, να επιμείνω για την ανάγκη να βρούμε τεχνικές λύσεις, για αυτές που αναφέραμε δηλαδή προηγουμένως. Η διαλειτουργικότητα είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο δεν χωρούν συμβασμοί, αλλά ούτε και καθυστερήσεις. Διαφορετικά διατρέχουμε τον κίνδυνο κερματισμού λόγω ακριβώς αυτής της έλλειψης διαλειτουργικότητας, κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά στη Σουηδία. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε επενδύσει, οι οποίε είναι απαραίτητε. Αν δεν γίνουν, διατρέχουμε κινδύνου σοβαρού. Επίση, θα ήθελα να αναφερθώ στου κανόνε για τι κρατικέ επιδοτήσει προ του εθνικού φορεί σιδηροδρόμων για να ξεπεράσουν αυτή την πρώτη φάση επενδύσεων που πρέπει να κάνει ο τομέας των σιδηροδρόμων για να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Επίσης έχουμε να κάνουμε και με την επικουρικότητα στις ε, προτάσεις της ε, Κομισιόν σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Συγκεκριμένα θα, θα ήθελα να πω ότι στα άρθρα 4 με 6 της πρότασης της Κομισιόν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το θέμα της επικουρικότητας. Επειδή αυτά συγκεκριμένα τα άρθρα σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία των διοικήσεών μας και των εθνικών αλλά και των τοπικών. Η παρεμβάση λοιπόν σε αυτές τις εθνικές διαδικασίες θα ήταν αρνητική όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν καθυστερήσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και θα μπορούσαν να υπάρξουν μάλιστα και προσφυγή στα δικαστήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος για την παρέμβασή σας. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μαλοντίνοβιτς. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Είσαστε από την ε, Σερβία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς. Yeah. Thank you. Thank you. This is Ευχαριστώ, ξέρετε, είναι η πρώτη μου φορά και δεν άψα το μικρόφωνο. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, για εμά η συμμετοχή εδώ είναι πολύ σημαντική για διάφορου λόγου επειδή καταρχάς βρισκόμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων για προσχώρηση, αλλά όπως ξέρετε έχουμε μια στρατηγική θέση σε τρεις σημαντικούς ε, διαδρόμους της Ευρώπης. Μεσόγειος, ο Ανατολικός Διάδρομος και ο Διάδρομος του Δούναβη. Η Σερβία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των απαραίτητων προδιαγραφών ε, στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Ε, έχουμε εμπλακεί και, στην, και στο δημοτολόγιο διασυνδεσιμότητας στα Βαλκάνια, κάτι το οποίο έχει μεγάλη τοπική και περιφερειακή σημασία, με στόχο να κάνουμε πιο έντονες τη συνεργασία στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας. Ε, έχουμε διαδρόμους που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου και αναμένουμε και το πρώτο τερματικό πολύμορφο μεταφορών στο Βελιγράδι φέτος, ώστε να έχουμε όλες τις μορφές ε, μεταφορών οι οποίες θα προωθηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές βεβαίως της, και τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σε επιθυμίσω ότι και εμείς έχουμε επικυρώσει την ε, συμφωνία από το τέλος του 2017, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών στην περιφέρεια μας. Ευχαριστώ. Κράστα δύο λεπτά, έτσι ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρεμβασή σας. Ο λόγος στον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας, τον κύριο Ρικέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ για τους θαυμάσιους τους συζητές θα μας εισηγήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πράγματα τα εξής. Έχουμε ένα εργαλείο, μια διευκόλυνση το συνδέοντα στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει μια, ένα επιχειρηματικό λειτουργικό κομμάτι και ένα κομμάτι συντονισμού όπου συμμετέχουν χώρες μέλη. Και αναφέρθηκε βέβαια προηγουμένως και υπήρξε αμφιβολία κατά πόσο η εμπλοκή αυτών των ε, χωρών γίνεται με τρόπο εταιρική σχέση. Γιατί βλέπουμε ότι όταν διαθέτουμε τεχνικά μέσα, νομικά μέσα, λειτουργικά μέσα, τότε τα πράγματα προχωρούν. Είναι βέβαια σαφές ότι η δυνατότητα κατανάλωσης, η δυνατότητα για δημιουργία προσταμής αξίας, συντονισμού σε επίπεδο διευρωπαϊκών ε, δικτύων με τη διευκόλυνση αυτή οδήγησε σε κάποιες αμφισβήτητες επιτυχίες. Κανείς δεν το αρνείται αυτό. Θα πρέπει ενδεχομένως βέβαια να παραμείνουμε πιστοί στο αρχικό πνεύμα. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε κάποιες απλουστεύσεις εκεί όπου υπάρχουν πολυπλοκότητες, ε, να δούμε τι γίνεται με τα λειτουργικά επιχειρησιακά μέσα και το συντονισμό. Νομίζω ότι όσο προχωρούν τα δίκτυα, τόσο πιο πολύ ε, θα είναι ορατό το τέλος και θα ήθελα να πω ότι η ευρωπαϊκή μέθοδος έχει αποδειχτεί αποτελεσματική με τον τρόπο λειτουργίας της και νομίζω ότι, Πρόεδρε, θα πρέπει να τονίσουμε ακριβώς την αποτελεσματικότητα αυτού του εργαλείου και δεν θα πρέπει βεβαίως να αναφερόμαστε ενδεχομένως σε κάποια επιμέρους εργαλεία, τα οποία ενδεχομένως παρουσιάζουν και να ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε και ο κύριος Δελγάδο. Έχετε το λόγο. Ναι. Γεια σας κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές από την Ισπανία θα ήθελα να σας μεταφέρω ένα μήνυμα για το οποίο συμφωνούμε για την αναμφισβήτητη αποτελεσματικότητα και επιτυχία της πολιτικής των ευρωπαϊκών δικτύων για την ίδια την Ευρώπη και την ενιαία αγορά με την μεταφορά ατόμων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών προς τον πληθυσμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό από την Ισπανία το υπογραμμίζουμε. Θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για την πρόθεση αυτών των δικτύων μεταφορών που συμβάλλουν στην διάρθρωση και στην ενταφική συνοχή. Από την Ισπανία δέρχονται δύο διαδρομοί, του Ατλαντικού και της Μεσογείου, που δέρχονται σε, από, 10, από τις 17 αυτόμες περιοχές. Θα θέλαμε η Κομισιόν λάβει υπόψη της την ισπανική πρόταση για διεύρυνση κάποιου από αυτούς τους διαδρόμους, πέραν δηλαδή του Μεσογειακού και του Ατλαντικού που εντάσσονται στο κανονισμό. Συγκεκριμένα έχουμε τις ε, διαδρομές Κορούνια Λεόν, Ουέλβα Σεβίλια, Παπλώνα Λογρόνιο, ε, Νότια πάλι Ισπανία Ανταλουσία και επίσης ο διάδρομος με τις Βαλιαρίδες και τα Κανάρια νησιά. Γιατί αυτοί οι διάδρομοι έχουν παραμείνει στο περιθώριο και θα πρέπει να ενισχυθούν. Ελπίζουμε τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να κάνουν τις απαραίτητες εγκρίσεις μέχρι το 2021. Θα ήθελα να τονίσω την σημασία προώθησης της συνδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων. Είμαστε πρωταθλητές στους επιβάτες, έχουμε όμως κάποια στέρηση στα εμπορεύματα και όπως ακούσαμε προηγουμένως για το Ρότερνταμ είναι απαραίτητο να προωθήσουμε τις συνδέσεις με τους λιμένες, δηλαδή είναι σημαντικό να έχουμε σύνδεση οδικών μεταφορών με λιμένες και τέλος να τονίσω την σημασία των συστημάτων διαχείρισης ε, κυκλοφορίας όπως το RMTS που έχει τεράστια σημασία και για τις υδρομικές μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντελγάδο. Ο κύριος Καματερός έχει το λόγο. Πού είσαστε κύριε Καματερέ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Μεταφορών. Έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ε, είπε ο κύριος ε, Γκρός για το πρόγραμμα, για το διάδρομο Orient East ε, στον οποίο συμμετέχει και η χώρα μας. Ε, όμως πρέπει να τονίσω ότι είναι το μοναδικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει. Και σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις του κανονισμού από αυτό το πρόγραμμα και εμείς βρισκόμαστε στη διαδικασία εκπόνησης εθνικού στρατηγικού σχεδίου μεταφορών ε, με ορίζοντα το 2037 και ενδιάμεσο χρονικό ορίζοντα το 2027. Ε, παράλληλα θεσμοθετούμε μέτρα όπως τα συστήματα ψηφιακών μητρών, ηλεκτρονικό εισιτήριο εφιών συστημάτων μεταφορών, ηλεκτρονικό σύστημα αναλογικής χρέωσης διοδίων και άλλα. Το έργο περιμένουμε να έχει ολοκληρωθεί, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2019 και φυσικά χρηματοδοτείται από κοινοτικά προγράμματα. Ε, όμως ε, η χώρα μας δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Η βελτίωση και η ανάπτυξή του θα στηρίζεται στις συνδυασμένε μεταφορές από αέρα ξηρά θάλασσα που πέραν του γενικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνει ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα ε, και λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της διαμόρφωσής της. Ε, να σας θυμίσω ή να σας τονίσω ότι ε, η χώρα μας αποτελεί τη φυσική πύλη προς την ε, Ευρώπη είναι ένα διεθνές διαμετακομιστικό ε, κέντρο, είναι ενεργειακός κόμβος, ε, πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός, είναι μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη ε, και θέλουμε, η πολιτική που ακολουθούμε είναι ότι θέλουμε το, τα Βαλκάνια γενικότερα και χαίρομαι πολύ που άκουσα και τη γειτόνισσα από τη Σερβία να είναι ένας, ένας παγκόσμιος επενδυτικός προορισμός να είναι ένας χώρος ειρήνης, σταθερότητας και ισότιμης συνεργασίας και δεν είναι τυχαία η συμφωνία που υπογράψαμε αυτέ τι μέρε ε, με την ε, γείτονά μα, ε, την Φύρομ. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαν Ντίκ ότι οι θαλάσσιες μεταφορές έτσι όπως φαίνεται και θα θέλαμε μία τοποθέτηση πάνω σε αυτό είναι λίγο είναι υποβαθμισμένες και όμως θα επεκτείνω ε, την, ε, το πρόβλημα αυτό και θα ζητούσα ε, να μην βλέπουμε μόνο τις μεταφορές εμπορευμάτων αλλά, και ανθρώπων και εδώ θα πρέπει να δούμε τη σχέση και με τον τουρισμό στην, μετα, στις θαλάσσιες μεταφορές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καματέρε. Ο κύριος Κράμερ, έχετε το λόγο για ένα δίλεπτο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Έχουμε, έχει αυξηθεί η κυκλοφορία γενικά στα δίχτυά μας. Ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να έχει προτεραιότητα. Είπαμε ότι 80% των χρημάτων πάνε στους σιδηροδρόμους. Αν δείτε όμως τα προγράμματα, βλέπετε που πάνε πραγματικά τα χρήματα. Κάνουμε πολλά σφάλματα στις επενδύσεις. Λοιπόν, βλέπουμε κάποια ποσά που δαπανώνται λάθος για τη διασύνδεση ε, Μπρεσλάου με Βερολίνο που κόστησε 100 εκατομμύρια διασύνδεση και κάποια σημεία δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί. Και ο διάδρομος από Κρακοβία σε Αμβούργο, αν ε, κατασκευαστεί, θα επιταχύνει πολύ τη διασύνδεση, αλλά δεν έχουν επενδυθεί σωστά τα χρήματα δίνονται δισεκατομμύρια για τα δίκτυα, αλλά είναι εμβαλωματικέ οι λύσεις και υπάρχουν κενά. κυρίω στα σύνορα υπάρχουν τα κενά, διότι δεν μπορούν να υποχρεώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη να εστιάσει σωστά για να ρίξει. Βλέπετε ότι υπάρχει κοινό 800 μέτρων στην Βαλενσιέν και θα μπορούσε μία ώρα να χρειαστεί για να γίνει το ταξίδι και δεν υπήρξαν χρήματα που διατάθηκαν για να συνδέσουν τη Γαλλία και την Γερμανία. Φράιμπουργκ με Κόλμαρ. Υπάρχει μία γέφυρα εκεί που καταστράφηκε πέρσι, κατέρευσε πέρσι και ακόμα η γέφυρα αυτή δεν έχει επιδιορθωθεί. Μόνο 5% των επιβατών που χρησιμοποιούν τους σιδηροδρόμους, χρησιμοποιούν τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Οι περισσότεροι επιβάτες χρησιμοποιούν μικρά ε, τοπικά τρένα. Αν δείτε τη Rail Baltica, είναι ένα, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, αλλά κοστίζει ελάχιστα σε σχέση με την γραμμή Λιών Τωρίνο. Δεν σημαίνει ότι είναι λάθος πρόγραμμα, αλλά χρειάζεται να φροντίσουμε τις διασυνοριακές διασύνδεσεις για να μπορεί να αναπτυχθεί σωστά η Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Συνεχίζουμε. Όχι, δεν χειροκροτούμε. Ακόμα και αν υπάρχουν εξαιρέσεις, ναι, ομολογώ, λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Κολακόσκι, Πολωνία. Καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η στήριξη του έργου της Επιτροπής σας όσον αφορά τις μεταφορές δηλαδή, είναι κάτι που βρίσκουμε πολύ καλό. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κάνετε υπέρ των προγραμμάτων υποδομών μεταφορών για τη σύνδεση των πρωτευουσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επόμενο πάντως μεγάλο σχέδιο στο οποίο θέλω να πιστήσω την προσοχή σας και όλων των Ευρωβουλευτών είναι ο άξονας που συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Ευρώπη. Θέλω να αναφερθώ στον ε, διάδρομο των Καρπαθίων. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει διαμετακομιστικές οδούς και θα μπορούσε να φροντίσει για τη σύνδεση των Βαλκανίων με τις Βαλτικές χώρες. Έτσι θα βοηθούσε και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, γύρω από τον Δούναβη για να συνδεθούν με τις υπόλοιπες χώρες. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσέγγισης που θα μπορούσε να συνδέσει πραγματικά όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και να φροντίσει για την ανάπτυξή τους. Θα έπρεπε να ενισχυθούν οι υποδομές εκεί υπέρ της ανάπτυξης και του εμπορίου μεταξύ της Ανατολικής Ευρώπης και της υπόλοιπης Ευρώπης ή και μεταξύ χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Σιδηρόδρομοι λοιπόν. Θέλω επίσης να πιστήσω την προσοχή σας σε ένα πρόγραμμα που ήταν υποψήφιο από πέρυσι, που είναι η συνδρομική σύνδεση υψηλή ταχύτητα από το Ταλίν μέσω της Πολωνίας μέχρι την Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα αυτό, με σχέδια υποδομών σε όλες αυτές τις χώρες, συνδρομικών υποδομών βέβαια. Αυτή η ταχεία σύνδεση είναι αναγκαία γιατί θα ένωνε το ανατολικό τμήμα με το βορρά και το νότο. Θα δημιουργούσε θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη, σταθερότητα σε αυτές τις περιοχές. Και θα και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ανατολικό τμήμα. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την ζημιά που υπέστησαν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μέχρι πρόσφατα, αξίζουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ τη δικιά σας στήριξη. Ο κύριος Γιαλούνεν. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ στην Επιτροπή σας. Μας θυμόσαστε, είχαμε, πάει στη... είχαμε έρθει στην ε, Φιλανδία και είχαμε βρεθεί, μας θυμόσαστε. Ωραία, καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο. Συγγνώμη, δεν σας άκουγα, λέει ο κύριος Γιάλωνεν. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, το θέμα ε, της ε, σύνδεσης με τη Βαλτική είναι κάτι σημαντικό και για τη Φιλανδία. Το ακούσαμε και πριν. Θα έπρεπε να περνάει η διαδρομή αυτή και από το Ελσίνκι από το Τελίν να πηγαίνει στο Ελσίνκι και μετά να συνδέεται με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της Φιλανδίας. Έτσι, μέσω αυτής της διαδρομής και στη Βαλτική μπορούμε να φτάσουμε και στην Ασία. Είναι γνωστή αυτή η σύνδεση μέσω Βαλτικής με την Ασία. Τώρα λοιπόν και σιδηροδρομικά θα έπρεπε να είχαμε κάτι αντίστοιχο. Στη Φιλανδία είναι δυνατόν να βρεθούν χρήματα για οδικές μεταφορές. Και θα έλεγα ότι σε χώρες όπως η Φιλανδία, όπου δεν υπάρχει στήριξη, θα έπρεπε να υπάρχουν ε, κίνητρα για επενδύσεις στις υποδομές. Κάτι το οποίο θα βοηθούσε τέτοιου είδου προγράμματα και θα ήταν προς όφελος ολόκληρης της Ευρώπης. Προτείνω λοιπόν να μιλήσουμε για διαφορετικές μορφές στήριξης εξαιτίας της επιτάχυνσης που δημιουργείται. Αλλά συγχρόνως επιτρέψτε μου και να σας υπενθυμίσω ότι δεν μιλάμε για τις παραδοσιακές μεταφορές, ούτε καν τις γιατί υπάρχει νέα τεχνολογία, υπάρχουν εξελίξεις τεχνολογικές ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και σίγουρα στο μέλλον θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε ακόμα και drones ενδεχομένω. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, ότι υπάρχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες ο εχμής, όποτε μιλάμε για τις μεταφορές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Λαυστρόμ. Πού είσαστε? Α, εκεί. Ωραία. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε αυτοί που θα κερδίσουν στην, ε, στις μεταφορές και στην αυσιπλοεία πιο συγκεκριμένα είναι αυτοί που θα χρησιμοποιήσουν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Με αυτές που συνεισφέρουν σε χαμηλές εκπομπές και σε πιο αποτελεσματική χρήση των σκαφών. Το LNG ε, εισήχθη στη Φιλανδία ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε ε, το θέμα των καυσίμων. Η συμμετοχή τώρα των δρόμο της θάλασσας είναι κάτι σημαντικό και για μας. Και το σχέδιο αυτό ελπίζω να συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο και να έχει χρηματοδότηση. Στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να υπάρξει αύξηση των κονδυλίων για την έρευνα και την ανάπτυξη υπέρ ακριβώ τη ναυσιπλοεία, ώστε να εκπέμπει όσο γίνεται λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Αλλά βέβαια και η υλοποίηση, όπως είπε και ο κ. Φαντάκη, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Χρειάζονται πιλωτικά προγράμματα και δοκιμές, όπου βέβαια εκεί τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ της απασχόλησης, κάτι το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη για να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην ναυσιπλοεία με σκάφη ε, προηγμένης τεχνολογίας και αντίστοιχε υποδομές. Πρέπει συγχρόνω να αναγνωρίσουμε ότι η πραγματικότητα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στη Βαλτική θάλασσα ε, είναι πιο βαθιά τα νετά, τα ύδατα, με λιγότερο αλάτι. Είναι εντελώ διαφορετικά τα συστήματα που λειτουργούν. Η Φιλανδία έχει λιμάνια τα οποία παραμένουν παγωμένα 100 μέρες το χρόνο τουλάχιστον. Οπότε χρειαζόμαστε πιο βαριά σκάφη με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά για να υπάρχει ασφάλεια στην πλοία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι καταναλώνουν και περισσότερα καύσιμα και άρα είναι πιο ζημιογόνα για το περιβάλλον. Η ναυσιπλοεία λοιπόν στον πάγο είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να τιμωρούμε μία περιοχή της Ευρώπης βάζοντας κριτήρια που είναι καλά για λουπ. Ευχαριστούμε πολύ. με κυρία Ντεμόντε έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές για τις εισηγήσεις τους και τις πληροφορίες που μας έδωσαν ώστε εμείς να είμαστε σε θέση να σχηματίσουμε άποψη και να συζητήσουμε πολιτικά. Σήμερα καταγράφω, πρέπει να πω με κάποια απογοήτευση, ότι έχουμε τον κύριο Ιμπανέ, Ιμπανέζ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο κυριότερος αντίπαλος της γραμμής Τωρίνο Λιών και ο πιο μεγάλος πολέμιος. Μάλιστα σε σημείο που ήρθε σε σύγκρουση με τις τοπικές κοινωνίες του Τωρίνο και της λιόν. Ελπίζω να διαψευστώ και να μην είναι έτσι. Αν λοιπόν πρέπει να κάνουμε συζήτηση πολιτική, πρέπει να έχουμε ισορροπέ θέσει. Αν κάποιο αναφέρθηκε αρνητικά, πρέπει κάποιο να μιλήσει και αντίστροφα. Αλλιώ η συζήτηση είναι εκτό τόπου. Οπότε, ερώτηση προ εσά για διευκρινήσει. Θα θέλατε να μα πείτε ποια είναι η εναλλακτική που βλέπετε σε σχέση με αυτή την γραμμή. Σα παρακαλώ όμω να μου δώσετε μια άποψη όχι ακτιβιστή, αλλά οικονομολόγου. Δεύτερη ερώτηση για τον κύριο Κρότ για τα Βαλκάνια. Έχουμε αυτό το νέο στοιχείο για την κοινότητα μεταφορών. Θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς ποιες συγκεκριμένες προοπτικές υπάρχουν, τι δυσκολίες υπάρχουν και κάτι άλλο ως πληροφορία που θα ήθελα από εσά είναι να μου πείτε αν υπάρχουν κινέζικες επενδύσεις εδώ και πώς ακριβώς εμφανίζονται, ποια μορφή έχουν αυτές οι κινέζικες επενδύσεις στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντελμόντερ. Τελευταίο αλλά όχι λίγο το σημαντικό, ο κύριος Τελίνσκα. Έχετε το λόγο. Βλέπω ότι είσαστε, έχετε καλή διάθεση. Αστείευεστε, με πειράζετε. Δεν είναι απλώς ακρόαση, αλλά ε, και ερχόμαστε σε επαφή με του συναδέλφου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Λοιπόν, κάποιε αντιδράσει και μια έκκληση έχω. Πρώτα απ' όλα, προς τον Λετωνό συνάδελφο να πω, η Rail Baltic, η Rail Baltic έχει προτεραιότητα δικαιολογείται, διότι σημειώνεται πρόοδο. Είμαι πρώην Ευρωπαίο συντονιστή για αυτό το θέμα και χαίρομαι που ακούω ένα λετωνό πολιτικό που είναι τόσο θετικό και ενθουσιώδης. Για εσά από τη Ρουμανία, κύριε Μπόρθουμ, δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ Ανατολική Ευρώπη με Κεντρική Ευρώπη και Δυτική Ευρώπη. Έχουμε ενιαία αγορά, έχουμε προτεραιότητε και σχετικά με αυτό είμαστε συνδεδεμένοι και αυτό είναι ο ρόλος της διασυνδεσιμότητας μεταξύ μας. Θα έχετε το μερτικό σας, αλλά πρέπει να το εξετάσουμε. Είναι περίπλοκο το θέμα. Προς συναδέλφου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μια σχόλια, ένα από του δύο εισηγητέ για το ΣΕΦ, για το Μέσο σύνδεση τη Ευρώπης. Εάν μπορούσατε να μας δώσετε δικές σας ιδέες, Αυτό το Connecting Europe Facility, αυτό το μέσο για τη σύνδεση της Ευρώπη. Ε, πού βλέπετε ότι κάτι του λείπει σε εθνικό επίπεδο να παίξετε ένα ρόλο, τα εθνικά κοινοβούλια να παίξετε ένα ρόλο. Είναι αρκετά ε, περίπλοκα προβλήματα και αποτελματώσεις σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά το πάνελ, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το ΣΕΦ, όλα αυτά έχουν πετύχει. Μία αίτηση έχω. Από πλευρά του κ. Βαντάικ. Έβαλε συστάσεις για το ΣΕΦ 2. Οι υπόλοιποι όμως λένε Κάτι θα ήθελα να μου πείτε τι λείπει, τι θα έπρεπε να καλυφθεί και δεν καλύπτεται. Ο Μάτιο Γκρός είναι σε πολύ καλή θέση, σαν Ευρωπαίος συντονιστής για αυτά. Προς τον κύριο Βαντάικ, το blending, αυτή την ανάμιξη, το blending, πώς το αντιλαμβάνεστε, σαν λιμάνι. Το λιμάνι εξορισμού είναι κερδοφόρο. Το blending για κέρδος πώς λειτουργεί και μετά βλέπουμε και ποιος είναι ο ρόλος αυτής της ανάμειξης, το blending. Τέλος, σχόλιο. Κάποιος αναφέρθηκε στην ημερομηνία του 64. 60-40. Νέα ανάπτυξη, εξυγχρονισμός. Αυτό είναι σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στο λιμάνι σας όμως τι ισχύει. Θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη απλούστευση, ναι ή όχι. Αυτή είναι μια από τι ερωτήσει και σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τελίνσκα. Σημαντικά θέματα, σημαντικέ ερωτήσει. Θα έχετε ελάχιστο χρόνο. Λυπούμε γι' αυτό. Αλλά είστε λακωνικοί και θα έχετε ένα δίλεπτο ο καθένας. Λακωνικοί και περιεκτικοί. Θα ξεκινήσουμε όπως πριν. Κύριε Κόλσον, πρώτος. Θυματάρχη στη DG Move. Σας δίνω το λόγο για δύο λεπτά και ξεκινάω το χρονόμετρο από τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά σε κάποιες. Καταρχάς τον κύριο Ρικέ. Πράγματι στο ΣΕΦ υπάρχει πρόγραμμα που προσπαθεί να ενισχύσει το ρόλο του συντονιστού, να δημιουργήσει περισσότερες σχέσεις μεταξύ επιλογής προγραμμάτων που από το ΣΕΦ και του ρόλου του συντονιστού. Και αυτό ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Δεύτερο στοιχείο. Αυτή η αντιπαράθεση που καμιά φορά βλέπουμε μεταξύ μικρών και μεγάλων προγραμμάτων. Δεν υπάρχει τέτοια αντιπαράθεση. Έχουμε τους διαδρόμους που διαχειρίζονται πάρα πολύ ε, μεγάλη κυκλοφορία. Χρειάζονται μεγάλα προγράμματα. Δεν σημαίνει ότι, ότι θα πρέπει να αφήσουμε εκτό τα μικρά προγράμματα. Το Rail Baltica είναι ένα πρόγραμμα πολύ θεμελιώδες όσον αφορά τι μεταφορές, είναι για στρατηγικά σημαντικό και για να συνδεθούν τα βαλτικά, οι χώρες με την Ευρώπη και του πολίτε Ευρώπη. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα είναι ε, σοβαρό σφάλμα. Όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Δελμόντε για, το, για τη σύνδεση Λιών-Τωρίνο. Εγώ δεν θέλω να αντιταχθώ σε κάποιον προλαλήσαντα. Να πω ότι δεν συμμεριζόμαστε εμείς τη δική του θέση. Είναι σαφέστατο. Πρώτα απ' όλα η παρούσα γραμμή είναι ανίκανη να αντέξει επαρκή κυκλοφορία σε ένα διάδρομο όπως είναι ο διάδρομος της Μεσογείου. Είναι ξεκάθαρο λόγω του ευρου από τι ράγε, λόγω των, κλίσεω κλπ. Θα μπορούσα να αναφέρω διάφορε λεπτομέρειε επί ώρε. Μετά το κόστος του προγράμματος δεν είναι αυτό που αναφέρεται. Είναι πιο μικρό το κόστος, ακόμα προσθέτοντας και διάφορα, διάφορες λεπτομέρειες. 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Λιγότερο λοιπόν από αυτό που αναφέρθηκε. Τρίτο στοιχείο. Το μεγάλο λάθος που κάνουν κάποιοι που είναι αντίθετοι είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η Λιόν ε, του Ορίνου δεν είναι ένα πρόγραμμα μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, Λιών και του Ορίνου. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα για ένα διάδρομο που αντιπροσωπεύει έναν όγκο τεράστιο ε, ροών. Ευχαριστώ, κυρία Κόλσον. Κύριε Ρος, εσείς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε για τη Λιόν Τωρίνο, να πω το εξή. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των διευρωπαϊκών δικτύων είναι που κινείται προς τον ορίζοντα 2030 και προστατεύεται από τις συζητήσεις εθνικού επίπεδου στιγμίας φύσεως. Τώρα, αν είναι καλά βάσιμο το πρόγραμμα ή όχι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είδα στους διαδρόμους σε κάποιες χώρες που έχουν αλλάξει άπειρες κυβερνήσεις και δεν άλλαξαν ποτέ προτεραιότητες ε, όπως γι' αυτό είχαμε την επιτυχία στην Ελλάδα και τις επενδύσεις που είδαμε όταν κάναμε επίσκεψη στην Ελλάδα πριν από δύο-τρει εβδομάδες. Τώρα όσον αφορά τις επενδύσεις μας, πρέπει και αύριο να δούμε τι προστιθέμενη αξία δίνουν για εκείνου που ζουν κατά μήκο των διαδρόμων. Μια συνεργασία ενισχυμένη με τα διεθντικά ταμεία είναι κάτι σημαντικό. Δεν είναι ουσιαστικό κυριστικό να συνδέσουμε το α με το β, αν δεν ασχοληθούμε με αυτούς που ζουν μεταξύ α και β. Και εκεί τα διαθωτικά ταμεία που έχουν πολλά μέσα μπορούν να συνεργαστούν με το μέσο για τη σύνδεση της Ευρώπης, το ΣΕΦ, για να δώσουν προστιθέμενη αξία. Όσον αφορά τα Βαλκάνια, θα έλεγα όσον μας αφορά, ζητούμε δύο πράγματα. Να ακολουθηθεί μια λογική των εισαγωγικών σύνδεσης, να μην επενδύονται σε χώρες, σε μονόδρομους, σε διαδρόμους που υπάρχουν στην Ευρώπη και θα μπορούσαν να υπάρχουν αύριο μαζί τους να, να επικεντρωθούμε. Και δεύτερον, υφετηθούν ήδη κριτήρια, κριτήρια τεχνικά διαλειτουργικότητας ευρωπαϊκής, για να μην έχουμε αύριο προβλήματα τεχνικά, που είναι κάτι δαπανηρό, το εύρος από τις ράγες είναι κάτι σημαντικό και όσον αφορά τις κινέζικες επενδύσεις, προσωπική μου άποψη, πρέπει να το προσέξουμε, να προσέξουμε τις κινέζικες επενδύσεις διότι κινδυνεύει να είναι φθηνό χρήμα, βραχυπρόθεσμα, πολύ βραχυπρόθεσμα, αλλά που θα είναι πολύ ακριβό αύριο. Πιστεύω ότι εκείνοι που χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα θα πρέπει να σκεφτούν μια στατηγική μακροπρόθεσμη και όχι χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμη. Σαν συντονιστές δεν έχουμε άλλη φιλοσοφία να εξηγήσουμε. Από εμπειρία μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιε περιφέρειες που βλέπουν την ποιότητα τη δουλειά που γίνεται βάσει ευρωπαϊκών κριτηρίων και την ποιότητα τη δουλειά που κάνουν άλλοι. Όσον αφορά την Ελλάδα, επανέρχομαι σε αυτό, είναι ένα παράδειγμα η Ελλάδα συνέχεια όσον αφορά θετικών επενδύσεων. Κάτι που προβλέπουμε για το μέλλον. Με μια συνεργασία από τα ιδιωτικά ταμεία που είπα πριν, μπορούμε έτσι πραγματικά να αυξήσουμε ήδη την αξία των επενδύσεων που ήδη έχουν γίνει εκεί. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκρός. Όχι, ο κύριος Συμπανές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόλσον νομίζω ότι έκανε πραγματικότητα την ευχή σας. Είδατε ότι η Γενική Διεύθυνση MOVE εξήγησε ότι δεν είμαστε πάντα σε θέση να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Στα 1500 μέτρα ύψος οι Ελβετοί, στα 1600 οι Αυστριακοί κλπ. Είδατε ότι μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν ε, πολυτροπικές μεταφορές. Η απάντηση είναι πολύ βασική. 120 τρένα υπήρχαν τη δεκαετία του 80 με μία γραμμή. Τώρα 20 την ημέρα. Αν κάνουμε όπως τη δεκαετία του 80 και σήμερα, με 28 βαγόνια. Αν πολυπλασιάσετε όλε τι μέρε κτλ., φτάνουμε σε 980 τόσε χιλιάδε, δηλαδή 75% των ε, βαγονιών στο δρόμο. Είναι μάθημα βασική οικονομία, έτσι, αρκεί να κάνει κανεί πολυπλασιασμού και προσθέσει. Ένα πράγμα έχω να σα πω. Οι πολιτικοί σα φίλοι συνέταξαν συμφωνίε ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία. Το θέμα δεν είναι ούτε της Γαλλίας που σταμάτησε τον Ιούλιο 17, ούτε Ιταλίας που είπε ότι θέλει να ξανασυζητήσει το σχέδιο εφαρμόζοντας τις συνθήκες. Δεν λέμε σταματάμε, λέμε εφαρμόζουμε τη συνθήκη που οι δικοί σας φίλοι συνέταξαν. Και τι λέει η συνθήκη, τι λέει η συμφωνία, ότι η Γαλλία δεσμεύεται να πληρώσει 5 δισεκατομμύρια παραπάνω στις γαλλικές υποδομές από ό,τι η Ιταλία. Και γι' αυτό οι Ιταλοί πληρώνουν περισσότερο. Τώρα αν οι Ιταλοί θέλουν να πληρώσουν περισσότερα για το διασυνοριακό τούνελ χωρίς αντιστάθμισμα από την γαλλική πλευρά, εντάξει, μπράβο, εξηγήστε το όμως και στους ψηφοφόρους σας. Τελικά όλα αυτά είναι βασικές αρχές οικονομίας. Όσον αφορά τους ακτιβιστές, γιατί έτσι με αποκαλέσατε, επιτρέψτε μου να σας δείξω αυτό. Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες της Γαλλίας, όλη η γαλλική διοίκηση, το Γενικό Συμβούλιο για τα οδοστρώματα κτλ. Το Συμβούλιο Οικονομικών, η Διεύθυνση του Εσωβροφικυλίου, το Ελεκτικό Συνέδριο κλπ. Όλοι αυτοί είπαν ότι το σχέδιο αυτό δεν είναι οικονομικά συμφέρον. Μπορείτε να συνεχίσετε να λέτε ό,τι θέλετε, κυρία Πρόεδρε, αλλά οι οικονομολόγοι δεν είναι ακτιβιστές, είναι η κεντρική γαλλική δίκαιση. Και αυτό που είναι περίεργο είναι ότι εδώ και 20 χρόνια Όλες αυτές οι πληροφορίες, όλα αυτά τα συμπεράσματα αγνοήθηκαν τόσο από την ευρωπαϊκή κοινότητα όσο και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ισχύει αυτό πια, ευτυχώς το καλύτερο. Με τη σημερινή κυβέρνηση, με την Υπουργό Μεταφορών στη Γαλλία, με αυτόν που και αντίστοιχα Υπουργό στην Ιταλία, πρέπει να γίνει πραγματική συζήτηση. Και ναι, η υπάρχουσα γραμμή μπορεί να βγάλει ένα εκατομμύριο φορτηγά, το 70% όπως ζήτησε πριν και ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστούμε κύριε Παύλεφ. Κύριε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Να σχολιάσω περισσότερο κάποια σημεία που αναφέρθηκαν. Είχαμε από το ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ κάποια ποσά, κάποια δισεκατομμύρια δηλαδή για τις υποδομές και την εφαρμογή αυτών των έργων, την υλοποίησή τους. Τώρα θα πρέπει να δούμε και την αναλογία μεταξύ τους. Μήπως θα πρέπει ας πούμε να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων και στην εφαρμογή τους σε σχέση με το ευρύτερο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και είχαμε μια έρευνα τα τελευταία πέντε χρόνια που έδειχνε ότι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό πήγε στα λιμάνια, στους λιμένες και βλέπουμε πια ότι αυτά τα έργα για τους λιμένες δεν είναι πια κάτι το θεωρείται πια κάτι το τοπικό είναι υποδομές οι οποίες έχουν μεγάλο διασυνοριακό αντίκτυπο οπότε μέσω των λιμενών μπορούμε ας πούμε να προωθήσουμε τη μεταφορά εμπορευμάτων τη σιδηροδρομική να κάνουμε διασυνδέσεις μεταξύ διαφόρων ε, σημείων ενδιαφέροντος προς το εσωτερικό της χώρας κτλ. Αυτό περιλαμβάνουν πια διάφορα έργα και με αυτή την οπτική γωνιά θα πρέπει να κρυθούν. Επιπλέον να πω ότι για τα λιμάνια βεβαίως θα συμφωνήσουμε. Ε, είχαμε και ένα έτος διαπραγματεύσεων με τα εθνικά κοινοβούλια για εξυγχρονισμό και αυτό είναι και κάτι πια που νομίζω ότι οι λιμενικές αρχές το δέχονται, το αποδέχονται και βλέπουν και οι ίδιες τις προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα των, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης. Οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώς εδώ τι γίνεται με αυτό το 60 και το πώς υλοποιείται. Μετά για τον συνδυασμό, το blending για το κατά πόσο ας πούμε εμείς είμαστε κερδοφόροι και νομίζω ότι όντω είμαστε κερδοφόροι αυτό διαφαίνεται και από, τις, από τους λογαριασμούς μας τώρα έχουμε και ένα νέο κανονισμό που έχει υιοθετηθεί και ελπίζω σε δύο-τρία χρόνια θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια για να δούμε πιο ξεκάθαρα όλα, όλα αυτά τα στοιχεία γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ε, διαφάνεια Επαναλαμβάνω λοιπόν, ναι, είμαστε κερδοφόροι ως λιμένας του Ρότερνταμ και επανεπενδύουμε στον ίδιο τον λιμένα. Τώρα, μήπως θέλετε παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Είχαμε 306 ε, εκατομμύρια ε, έργο, 6 από επιδοτήσεις κρατικές και πολύ περισσότερες από το ίδιο το λιμένα. Ε, τα συνδυάζουμε όλα αυτά με τρόπο νομίζω αποτελεσματικό. Αν θα δείτε και ε, τα επιτόκια με τα οποία δανειζόμαστε είναι πάρα πολύ καλά στην αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρος. Σας παρακαλώ, μάλλον σας καλώ να χειροκροτήσουμε τους ηγητές μας για τις ποιοτικέ τους εισηγήσεις. Ουσιώδη ζητήματα προσεγγίσαμε για τη χρηματοδότηση των υποδομών νομίζω έχουμε πια διαφορετική οπτική και αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τις επιλογές με διαφορετικό μάτι. Λαμβάνοντας υπόψη το θέμα διαφάνειας καταρχάς. γιατί όλα αυτά που κάνουμε αφορούν τους πολίτες, τους άντρες και τις γυναίκες της Ευρώπης και την καθημερινή τους ζωή. Και ένα θέμα που αναφέρθηκε πολύ σημαντικό ο κύριος Δελγάδο το έθιξε λέγοντας ότι κοιτάξτε τα φορτηγά στα τρένα είναι προτεραιότητά μας. Υπάρχει η κλιματική αλλαγή και όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι και θα έχουμε πρόβλημα αν δεν μειώσουμε σημαντικά τους δρύπους διοξιδίου άνθρακα μετά από τη Συμφωνία του Παρισιού. Τώρα πια οι μεταφορές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και την ευθύνη που έχουν και να την αναλαμβάνουν και ξέρετε ότι ακόμα απέχουμε πολύ από αυτό. Οπότε θα πρέπει να επιταχύνουμε τον ρυθμό μας, γιατί δεν δουλεύουμε μόνο για μας, δουλεύουμε για τις μελλοντικέ γενιές και για το μέλλον του πλανήτη μας. Επίσης πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες δομές. Μιλήσαμε για το Λιόν, το Ρήνο. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν έργα τα οποία είναι προβληματικά. Είναι προβληματικά επειδή δεν συζητάμε για αυτά τα θέματα. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλα τα μέρη να συζητήσουν, να κάτσουν να συζητήσουν όχι με μια προοπτική πενταετίας, δεκαετίας, αλλά δεκαπενταετίας. Γιατί οι υποδομές δεν εξαντλώνται σε προεκλογικές εκστρατείες. Έχουν μια προοπτική μέλλοντος και μακρόπνοη μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς, κύριοι, και λέω κύριοι γιατί είμαι μόνη γυναίκα εδώ, θα ήθελα σας παρακαλώ να αποχωρήσετε από τις θέσεις και να τις παραχωρήσετε στους επόμενους ομιλητές. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εισηγήσεις σας. Έχουμε τη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα, η οποία θα ασχοληθεί θα ασχοληθεί με τις προοπτικές και τις προκλήσεις μετά το 2020 όσον αφορά την χρηματοδότηση των υποδομών στον τομέα των μεταφορών. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ολολάη, από τον Γενικό Διευθυντή της MOVE, της, από την Κομισιόν, να έρθει να καθίσει εδώ. Monsieur Dunet, qui est le directeur du... Κύριος Διευθυντή για θέματα κινητικότητας. Α, κάνετε πολύ φασαρία, λέει πρόεδρο. Σας παρακαλώ, αν θέλετε να μιλήσετε, να βγείτε έξω. Από την Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων, λοιπόν, κ. Δενέτ, υπεύθυνο θεμάτων κινητικότητας. Σας παρακαλώ, βγείτε έξω σιγά σιγά και ο κύριος Brian Simpson, Ευρωπαίος Συντονιστής των Θαλασσίων Διαδρομών, Θαλασσίων Οδών. Χωρίς να χάσουμε λοιπόν χρόνο, θα δώσω το λόγο κατευθείαν στον κύριο Λολάη, Γενικό Διευθυντή της ΜΟΥΒ και συνάδελφοι Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας παρακαλώ να συμμετάσχετε στη συζήτηση αλλά για να το κάνετε αυτό βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το πορτοκαλί δελτίο αν έχετε ερωτήσεις που θέλετε να θέσετε. Παρακαλώ ησυχία, ησυχία, ησυχία. Όσοι θέλετε να μιλήσετε να βγείτε έξω. Ξεκινάμε λοιπόν. Αν έχετε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια ερωτήσεις, αρκεί να συμπληρώσετε αυτό το πορτοκαλί δελτίο. Και ρολάει Ξεκινάτε εσείς, έχετε το λόγο από την κυρία Διευθύνση Move, έχετε 7 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι εδώ και έχω με χαρά αυτή την ευκαιρία κυρίες και κύριοι να σας μιλήσω για τη χρηματοδότηση των υποδομών. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι κέριο αυτό που κάνουμε σήμερα, που συζητάμε, μετά από την πρόσφατη υιοθέτηση της πρώτης της Κομισιόν για τη χρηματοδότηση των μεταφορών υπό το νέο μακρόπνο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Έχουμε λοιπόν ανάγκες χρηματοδότησης 500 δις από το 21 μέχρι το 30 σε σχέση με τα δίκτυα που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. 1,5-3 συνολική χρηματοδότηση των υποδομών μεταφορών συμπεριλαμβανομένων όλων των δικτύων και αν θέλουμε πραγματικά να επιταχύνουμε την μετάβαση στην ευφυή e κινητικότητα στις αστικές περιοχές θα χρειαστούν περισσότερα κονδύλια. Το 2016 ήταν 1,8% χρηματοδότηση υποχώρησε από το 2002 το 2009. Είχαμε βέβαια την κρίση εντωμεταξύ. Οπότε έχουμε μία ανάκτηση σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά αυτό δεν επαρκεί ακόμα για τα χρόνια που είχαμε χάσει επενδύσεις. Οπότε έχουμε μια δύσκολη πρόκληση μπροστά μας. Πρώτη λοιπόν η Κομισιόν η υποδομή να συνεχίσει να χρηματοδοτείται πέραν του 2020 μέσω διαφόρων οικονομικών προγραμμάτων και εργαλείων. Αυτό ζήτησε η Κομισιόν. Αυτό δεν αφορά μόνο βέβαια τη διευκόλυνση σε στην Ευρώπη, αλλά και διάφορου ταμεία περιφερειακά, εδαφική συνοχή, ε, το όρος 2020, το επενδύοντα στην Ευρώπη κτλ. Το ΕΦΣΥ. Αυτό για να έχουμε υψηλής αποδοτικότητας υποδομή που θα συνδέει την Ευρώπη και όλες τις περιοχές της με τρόπο σύγχρονο, αποτελεσματικό, ασφαλή και βιώσιμο με απτά αποτελέσματα και ωφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν επίσης να τονίσουμε ότι χωρίς τους ιδιώτες οι εθνικές αρχές έχουν ανεπαρκή κίνητρα και πόσο μάλλον πόρους ακριβώς για να κάνουν αυτά τα έργα τα οποία έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντα λειτουργικά συστήματα και υποδομέ. Γι' αυτό ακριβώ θέλουμε να επικεντρώσουμε αυτή τη χρηματοδότηση τη κοινοτική σε υποδομέ υψηλή προστάμενη αξία και με περαιτέρω μόχλευση από άλλε πηγέ, συμπεριλαμβανομένου και του ιδιωτικού τομέα. Οπότε, τα διασυνοριακές ε, και η δυσονομική κρίση, κρίκη συγγνώμη, δεν έχουν αξιοποιηθεί. Γι' αυτό ακριβώ αυτό το εργαλείο διευκόλυνση, το συνδέοντα στην Ευρώπη, έχει εδώ σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να αναφέρω και άλλα δύο σημεία. Το 14-20 και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Είχαμε 23,2 τα οποία έχουν εγγραφεί στο υπεροπολογισμό για 643 έργα, τα οποία αναμένεται να κινητοποιήσουν 46,7 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικών επενδύσεων στην Ευρώπη. 96% του διαθέσιμου προπολογισμού έχει εγγραφεί, ε, κονδυλίων έχει εγγραφεί στο υπεροπολογισμό. Προωθούμε λοιπόν αυτά τα έργα προτεραιότητας με διασυνοριακή διάσταση και κάποια από αυτά είναι πολύ γνωστά που συνδέουν γνωστές περιοχές με υποδομή, τούνελ κτλ. Όλα αυτά τα κονδύλια ε, διαχειρίστηκαν στα πλαίσια του ΣΕΦ και ήδη η απόδοση αυτών των κονδυλίων αφορά το ίμιση της ε, περίοδου ως χρηματοδότηση. Πρέπει όμως να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιαστεί το εργαλείο. Η νέα πρόταση για το 2021-2027 προβλέπει σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αυτό οδήγησε την Κομισιόν υπό το τωρινό ΣΕΦ να υποβάλει σημαντικές ε, πρωτοβουλίες για το ΣΕΦ 2. Για τις μεταφορές έχουμε 30,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τη συγκεκριμένη περίοδο και αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 30% σε σχέση με την τωρινή περίοδο. Εδώ θα ήθελα να τονίσω τη μεγάλη σημασία και την σημαντική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ μιας αποτελεσματικής ε, διασύνδεσης ευρωπαϊκής μέσω της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Είχαμε και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου της 1ης του Μαΐου φέτο φέτος σε σχέση με την χρήση και την αξιοποίηση αυτού του πυλώνα που αφορά τις μεταφορές. Το νέο ΣΕΦ λοιπόν θα αφορά 12,8 δις από τη συνοχή 2,8 και έχουμε 6,5 νέα δις ευρώ από το φάγκλος και της στρατιωτικής κινητικότητας. Σύμφωνα με την ε, δέσμευσή μα βέβαια για την συμφωνία του Παρισιού όπου θα, περιλαμ... θα περιλαμβάνω τουλάχιστον ένα τέρο των κονδυλίων τα οποία θα συμβάλλουν στην ε, μετρίαση των... Ε, του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής. Η στόχευσή μας λοιπόν παραμένει στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων με ιδιαίτερη προτεραιότητα στο διασυνοριακό τομέα και στους ελίβοντες κρίκους των διευρωπαϊκών δικτύων που θα πρέπει να ακολουθούμε μέχρι το 2030, ώστε να διασφαλίσουμε συνέχεια και να ολοκληρώσουμε τα υποεξέλιξη προγράμματα. Ταυτόχρονα η πρότασή μα δίνει ευρύτερη και ισχυρότερη έμφαση στον εξοχρονισμό των υποδομών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειές μα για την διαχείριση των συστημάτων ασφάλεια όπω ΣΕΖΑΡ και άλλα συστήματα. Έχουμε την ψηφιοποίηση η οποία και αυτή θα πρέπει να επικρατήσει σε όλους τους τομείς ώστε να αποτελέσει τον καταλήτη όσον αφορά την αυτοματοποίηση και την ολοκλήρωση για τα νέα μοντέλα κινητικότητα. Ταυτόχρονα θα πρέπει τα δίκτυα μα να είναι ασφαλέστερα και ανθεκτικότερα στι θεομηνίε. Τα μελλοντικά λοιπόν προγράμματα θα αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τι συνέργειε μεταξύ των υποδομών ενέργεια και μεταφορών. Ιδιαίτερα θα υπάρχει συγκεκριμένη στοχευμένη εστίαση σε ε, μορφές υποδομών που θα προβλέπουν εναλλακτικές, ε, εναλλακτικά καύσιμα. Αναφέρθηκα προηγουμένως και στη στρατιωτική κινητικότητα. Νέο στοιχείο, νέα συνιστόσα των προτάσεων όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Και αυτό θα προωθήσει την διτή χρήση των υποδομών, δηλαδή των υποδομών που θα είναι απαραίτητε για την στρατιωτική κινητικότητα, που θα βασίζεται όμω και στι πολιτικέ ανάγκε, ανάγκε των πολιτών. Ταυτόχρονα και για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, αυτά τα κονδύλια θα επιτρέψουν τη ταχεία ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων, ώστε να έχουμε την κατάλληλη μετακίνηση των στρατικών υποδομών και των στρατευμάτων. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις μεταφορές και τις δράσεις μας όσον αφορά τις πολιτικές άμυνα, άμυνας. Δύο λόγια για το επενδύοντας στην Ευρώπη. Έχουμε αυτό το νέο ταμείο με 11,5 δις ευρώ που αφορούν υποδομές βιώσιμων μεταφορών θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις υποεπενδύσεων και να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες αποτυχίες ή κενά στις επενδύσεις ανά χώρα για να προωθήσουμε και την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να αναπτύξουμε στόχους όπου θα συμμετέχουν και οι ιδιώτες και να συνδυάσουμε κονδύλια από ιδιωτικές τράπεζες ή από εθνικές ε, τράπεζες ανάπτυξης. Ήδη έχουμε αρκετή εμπειρία για το συνδυασμό, για το blending από όλε τι χώρε μέλη υπό την τωρινή διευκόλυνση, το συνδέοντας στην Ευρώπη και νομίζω ότι είχαμε πολλά επιτυχή παραδείγματα, οπότε θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε αυτή την εμπειρία που έχουμε σχηματίσει μέχρι τώρα. Να συνοψίσω και να καταλήξω. Θα αναστήσουμε λοιπόν τη μέγιστη μόχλευση για τα δημόσια κονδύλια. Θα ακολουθήσουμε μια σφαιρική γενική προσέγγιση βάση των αναγκών αυτών των έργων και θα πρέπει να προετοιμαστούμε βέβαια κατάλληλα ώστε να ξέρουμε πώς θα αναπτύξουμε αυτά τα προγράμματα με την κατάλληλη συνέχεια που αν δεν την έχουμε βέβαια θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα ποιοτικά ε, προγράμματα τα οποία θα αξιολογηθούν. Και βεβαίως ε, οι χώρες μέλη ήδη έχουν κατανοήσει νομίζω επαρκώς για το πώς ακριβώς υποβάλλουν πια και κατάλληλες προτάσεις. Για να είναι ισχυρή ένωση πρέπει να έχουμε αποτελεσματικές υποδομές και βασιζόμαστε εδώ στην στήριξη του Εθνικού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων για την βελτίωση των υποδομών στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, λέει ο κύριος Ρικέ, επανέλαβε την Προεδρία. Ο κύριος Ντενέκ τώρα, ο οποίος είναι διευθυντής για την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παρακαλώ, για 7 λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ όλους για την πρόσκλησή σας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει ευρωπαϊκά προγράμματα εδώ και 60 χρόνια. Να, κάποια νούμερα. Είμαστε ε, μία από τις πρώτες ε, τράπεζες, από τα πρώτα θεσμικά όργανα που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανήκει στις χώρες μέλη η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Ανήκει σε όλες τις χώρες μέλη και μόνο στις χώρες μέλη. σε ποιον πρέπει να κάνω νεύμα για να προχωρούν οι διαφάνειες, για να ξέρω. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν έλεγα ότι πέρυσι επενδύσαμε πάνω από 78,2 δισεκατομμύρια σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι από τα πιο σημαντικά και επιτυχή οικονομικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί. Γιατί κάπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαιο δημιούργησαν έναν ισολογισμό πάνω από 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οπότε όταν ε, ακούτε να μιλάει κανείς για ε, χρηματοπιστωτικά εργαλεία, να ξέρετε ότι η ΕΤΕ είναι ένα από τα πιο σημαντικά τέτοια εργαλεία. Ωραία. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν έχουμε αναπτύξει τα προϊόντα μας, χαρτοφυλάκια, που πάνε από το δανεισμό, που αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητές μας, στο μείγμα με διάφορα άλλα μέσα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και βέβαια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρνουμε σε πέρας και διάφορες εντολές που είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα προς τις χώρες μέλη ή προς ε, παράγοντες που προχωρούν με προγράμματα. Ε, αναφέρθηκε νωρίτερα κάτι σχετικό, μπορείτε να ξέρετε το Γιάσπερ στο πρόγραμμα ή το Κέντρο Πραγματογνωμοσύνης, το Έλενα επίσης. Όλες αυτές οι εντολές συμβουλευτικού χαρακτήρα συνεχίζονται και είναι σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων μας. Τώρα το Τιμήμα στήριξη των μεταφορών από την τράπεζα είναι περίπου 12 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο δανεισμός προς όλους τους τομείς, αλλά όλο και περισσότερο μισός από αυτό το δανεισμό πηγαίνει στους σιδηροδρόμους, είτε πρόκειται για την ε, ύπεθρο είτε για τις αστικές περιοχές. Αλλά υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες που στηρίζονται σε άλλες μορφές μεταφορών δηλαδή. Δανείζουμε και εκεί. Δύο λόγια τώρα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα έχετε ακούσει αυτό το περίφημο σχέδιο Juncker, το οποίο βέβαια ολοκληρώνεται, ήταν πάρα πολύ επιτυχές, επεκτάθηκε, αλλά η τράπεζα έδωσε περίπου 350 δισεκατομμύρια επιπλέον επενδύσεις ως μόχλευση επιπλέον της εγγύησης που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επεκτάθηκε λοιπόν και έχουμε νέο στόχο τώρα προκειμένου να δημιουργήσουμε 500 δισεκατομμύρια μόχλευση σε όλους τους τομείς. Οπότε και στις μεταφορές με 25 δισεκατομμύρια ε, επενδύσει που δημιουργήθηκαν στον τομέα των μεταφορών. Τώρα, στρεφόμενοι προς το μέλλον, υπάρχουν ε, πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ακόμα ο κλάδος των μεταφορών. Θα τα ξέρετε φυσικά όλοι εδώ. Η μεγαλύτερη όμως είναι η χρηματοδότηση ακριβώς. Ακούσαμε για τις συζητήσεις που γίνονται αν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση ή όχι. Γεγονός είναι ότι η Ευρώπη δεν επενδύει αρκετά τα τελευταία δέκα χρόνια στα δίκτυα της μεταφορών. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή η έλλειψη επενδύσεων συσσωρεύεται. Μπορεί να μην φαίνεται αυτό από την αρχή, από την πρώτη χρονιά, αλλά υπάρχει μια συσσόρευση στην έλλειψη επενδύσεων και κάποια στιγμή οδηγούμεθα σε κρίση. Και όχι μόνο στις νέες χώρες και στις παλιές και πρέπει να προσθεθεί αυτή η καθυστέρηση στις επενδύσεις ε, γενικότερα στο πρόβλημα χρηματοδότησης και πρέπει να προσθέσουμε και οτιδήποτε καινούριο προκύψει. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Πρέπει να βρεθούν οι πόροι. Πρέπει να δούμε πώς, που και πώ βέβαια θα δαπανηθούν αυτοί. Φαντάζομαι ότι όλοι εσείς θα ασχοληθείτε με αυτό τα επόμενα δύο χρόνια που βάζουμε τις προτεραιότητές μας, πώ ε, βασίζουμε τα κριτήριά μας. Στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, προβλέπεται από το καταστατικό μας να επενδύουμε σε παραγωγικά προϊόντα. Οικονομικά παραγωγικά προγράμματα. Πρέπει να έχουν την προτεραιότητα. Αυτά. Λοιπόν, αυτή ήταν η τελευταία διαφάνεια και από εκεί και πέρα προσλέπω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντονέτ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Μπράιαν Σίμψον που είναι ο Ευρωπαίος συντονιστής για τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας. Μπράιαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, που ήμουν μέλος και πρόεδρος αυτού του ενδόξου σώματος, πάντα υποστήριζα περισσότερες επενδύσεις όσον αφορά τις μεταφορικές υποδομές και πάντα με υποστήριζαν τα μέλη της Επιτροπής. Τώρα νομίζω ότι έχουμε τα εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά μας και για να πετύχουμε το στόχο μας με μια συνεκτική πολιτική διευρωπαϊκών δικτύων και με το ΣΕΦ αλλά το έργο είναι πολύ μεγάλο δυσχερές. Θα είδατε να κυκλοφορούν διάφορα νούμερα σχετικά με το τι απαιτείται μέχρι το 2030. Αναμφισβήτητα, το ΣΕΦ είναι αποτελεσματικό εργαλείο, μπορεί να πετύχει διάφορους στόχους. Υπήρξε επιτυχές ή ήταν αποτελεσματικό. Έχουμε προγράμματα που αποδίδουν μεγάλη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Αν προσθέσετε σε αυτό τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ από το προπολογισμό συνοχής, βλέπουμε ότι δρέπουμε καρπούς από το δέντρο των μεταφορικών υποδομών. Πρέπει τα επιτεύγματα να τα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση. Και το ΣΕΒ στις επόμενες δημοσιονομικές προπτικές θα είναι εξίσου σημαντικό σαν εργαλείο όπως και πριν. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε το ότι οι μεταφορές θα έχουν ένα δίκιο κομμάτι της πίτας, διότι χωρίς αυτή την υποστήριξη όλα τα όνειρά μας θα παραμείνουν όνειρα. Η πρόταση που θετήθηκε στις 6 Ιουνίου τρέχοντος έτους θα είναι 30 δισεκατομμύρια ευρώ και ξέρω ότι κάποιοι από εσά θεωρείται ότι αποτελούν περικοπή. Αλλά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι η συμφωνία επ' αυτές τις περιστάσεις είναι δίκαιη. Ω συντονιστή για τους αυτοκινητόδρομους της θάλασσας, θα περιμένετε ότι εγώ θα υπερασπιζόμουν τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτός ο τομέας επί μακρόν ήταν η, ε, δεν ήταν η νύμφη, ήταν ε, παράνυμφος όσον αφορά τις κατευθύνσεις και την πρικοδότηση. Αλλάζουν τα πράγματα όμω. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι ο θαλάσσιος τομέα όσον αφορά την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο σύνολό τη. Υγούμεθα, αναπτύσσοντας εναλλακτικά καύσιμα. Υγούμεθα, όσον αφορά τη διαχείριση των θαλασσίων μεταφορών. Υγούμεθα, όσον αφορά την ανάπτυξη σταθερού συνεκτικού ε, ρόλου στην αλυσίδα της επιμελητία και τη οργάνωση τα τελευταία τρία χρόνια δαπανίσαμε 380 εκατομμύρια ευρώ σε 47 προγράμματα. Θεωρώντας ότι έχουμε 341 λιμάνια που υποδιούνται στους κανονισμούς ΣΕΦ και TNT, 79 από αυτά είναι σε έναν από τους 9 διαδρόμους και αυτά τα λιμάνια παίζουν κρίσιμο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, γιατί οι θαλάσσιες μεταφορές παίρνουν μόνο 4% από χρηματοδότηση του ΣΕΦ. Σας το θέτω σε εσά ως μέλη. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Και το ΣΕΦ 2 θα είναι μια καλή αρχή για κάτι τέτοιο. Δώστε στις θαλάσσιες μεταφορές ένα δίκαιο μερίδιο των πόρων. Βέβαια, θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Κατά την άποψή μου, το σημαντικότερο θέμα που αντιμετωπίζει ο τομέας στη μεταβατική φάση μεταξύ του f 1 και του f 2 είναι τα εξή. Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, μια ενιαία θηρίδα, αν θέλετε, και να προετοιμαστεί ο θαλάσσιος τομέας για ε, την, το ανώτατο όριο για το θείο για το 2020. Χρειάζεται περαιτέρω ψηφιοποίηση και πρέπει να παρέχεται υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG στα λιμάνια, ώστε ο τομέας να μπορεί να συμμορφωθεί με τις προθεσμίες του 2025. Εν γέννη, πρέπει να εξασφαλίσουμε καλό επίπεδο επάρκειας. Και θα πρέπει οι αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας να ενταχθούν στα διευρωπαϊκά δίκτυα και μετά το 2030. Γι' αυτό θεωρούμε ότι μας χρειάζονται 5 δις ευρώ, τόσο θα κοστίσει. Λοιπόν, αγαπητά μέλη, Δώστε μας τα εργαλεία και πιστέψτε με, θα κάνουμε τη δουλειά μας. Υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει, αλλά όλοι οι συντονιστές μας προσπαθούν να το κάνουν αυτό να πετύχει. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας κατά το παρελθόν. Και εδώ ελπίζω ότι ο θαλάσσιος τομέας τελικά θα γίνει νύμφη και δεν θα είναι πλέον παράνυμφος. Ευχαριστώ, Μπράιν. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Βέβαια, έχουμε καθυστερήσει κάπως και αυτό έχει γίνει κανόνας. Παρακαλώ τους παρεμβαίνοντας να μιλήσουν για ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να, να διακοπούν οι εργασίες μας από την άφηξη του Επιτρόπου Έτιγκερ. και ίσως τελικά να διακοπεί η θα τον ρωτήσω. Ο κ. Ντελγκάδο από την Ισπανία έχει το λόγο. Κύριε Ντελγκάδο, για ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό και όχι παραπάνω. Ευχαριστώ. Είμαστε υπέρ της αύξησης των επιδετήσεων στην διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη που από το 2014 χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση έργων και θεωρούμε ότι αυτός ο νέος μηχανισμός θα πρέπει να πρικοδοτείται από επαρκή κονδύλια για την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών δικτύων μέχρι το 2030 που έχουν χαράξει οι χώρες μέλη και που έχουν στηρίξει το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την χρήση καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων για αυτό το δίκτυο για την Ισπανία έχουμε 50 δις, 10% περίπου του συνόλου των βασικών υποδομών και έχουμε και επιπλέον χρηματοδότηση από άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θα ήθελα επί την ευκαιρία να χαιρετήσω την εργασία που κάνει η Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων, όπως είπε και ένας από τους προλαλήσαντε. Και πράγματι νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις επενδύσεις στις, στους αυτοκινητοδρόμους, στις παράκτιες περιοχές. Έχουν τεράστια σημασία και στην Ισπανία θα καταβάλουμε σοβαρές προσπάθειες για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δελγκάδο. Ο κύριος Σένεκε από τη Δανία έχει το λόγο. Έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου, δυστυχώς δεν τον ακούν οι διερμηνείς. Okay. Øh, tak for det, Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι μας που ασχολούμεθα με τις υποδομές στην καθημερινή μας ζωή, γνωρίζουμε τις μεγάλες πιέσεις που δεχόμεθα. Χρειαζόμαστε επενδύσεις σε καλύτερους δρόμους, ταχύτερα τρένα, καλύτερους ε, διαδρόμους για τα ποδήλατα και άλλα πράγματα στις χώρες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από διασυνοριακές επενδύσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα. Για κάθε ξεχωριστή χώρα υπάρχουν πολλοί οικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται. Και πολύ συχνά, όπως ακούσαμε σήμερα, ο πληθυσμός είναι διστακτικός. Υπάρχουν και νομικές επιπλοκές, υπάρχουν περιβαλλοντικές νομοθεσίες που διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από νομικό σύστημα σε νομικό σύστημα. Άρα χρειάζεται κουράγιο, χρειάζονται ήρεμη πολιτική όσον αφορά τα διασυνοριακά έργα. Η εμπειρία μας δείχνει όμως ότι όταν εφαρμόζονται, όταν υλοποιούνται τα έργα, τα αποτελέσματα είναι έξοχα. Στη Δανία είχαμε έξοχα οικονομικά αποτελέσματα, πολιτιστικά αποτελέσματα, χρηματοπιστωτικά αποτελέσματα και δημογραφικά αποτελέσματα εκεί που αποφασίζει ο κόσμος να ζήσει. Είχαμε καλές εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από διασυνοριακά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από αυτό. Είναι καλή ιδέα, αλλά είναι αδύνατο να υλοποιηθούν αν δεν έχουμε υποστήριξη και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διασυνοριακά έργα τα οποία είναι χρήσιμα, που έχουν νόημα, που μειώνουν εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και βοηθούν ποικιλοτρόπως. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χολέλα βέβαια για την παρουσίασή του και βέβαια πάντα υπάρχει ο κίνδυνος έτσι όπως το παρουσιάζουμε να ξεπεραστούμε με την επιτυχία. Τώρα εγώ θα ήθελα να πω κάποια πράγματα που δεν είπα νωρίτερα. Ότι δηλαδή για το καινούργιο συνδέοντα στην Ευρώπη θα έπρεπε να μπορούμε να οργανώσουμε κάποια συνέργεια ώστε όχι όπως έγινε τις τελευταίες φορές να υπάρχει κατακαιρματισμός θα έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση δεδομένης ακριβώ της εμπειρία που είχαμε από το παρελθόν. Και ακριβώς γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες μπροστά μας. Η κινητικότητα για τον ηλεκτρισμό, οι εναλλακτικέ που χρειαζόμαστε. Η πρόκληση η τεράστια που έχουμε μπροστά μας είναι όντως οι υποδομές για να φορτίζουμε μπαταρίες, τα ηλεκτρικά οχήματα και τέτοια. Οπότε, στον κύριο Χωρή θέλω να πω ότι εντάξει, υπάρχει συνέργεια όντως και με τον ορίζοντα 2020 που έχει μεγάλη χρηματοδότηση και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάποια μορφή τέτοιας συνέργειας που να διαθέτει συνέχεια στο χρόνο. Τώρα για αυτά που είπε ο κύριος Στάνετ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η μεγάλη αυτή διάδρομη χρειάζονται προγράμματα τα οποία να ενώνουν και να προσθέτουν μια προστιθέμενη αξία σημαντική. Και αυτό πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας για να μην εξαφανιστεί δυνατότητα της σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων διαδρόμων. Θα υπάρξει τέλος χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση, πιο φιλόδοξη από ό,τι λέει η Επιτροπή. Για να δούμε. Μακάρι να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε, γιατί το Συμβούλιο πάντα κόβει τα ποσά. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα Σέντερ. Ο κύριος Καμαρός, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος ε, Σίμψον, ε, που είπε ότι πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό της, ε, επιδότησης, της χρηματοδότησης της θαλάσσιας μεταφορές. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια παρατήρηση. Ενώ έχουμε πολύ σωστούς ε, στόχους σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, παράδειγμα για την ε, εδαφική συνοχή, πολλές φορές τα μέτρα που παίρνουμε, οι κανονισμοί που βγάζουμε έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Γιατί δεν είναι σωστό να παίρνουμε μέτρα οριζόντια, αλλά πρέπει να βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και με βάση αυτές τις ιδιαιτερότητες να παίρνουμε μέτρα. Θα σας αναφέρω ένα ή δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα αν προλάβω. Παράδειγμα, στην ε, Ελλάδα έχουμε 6.000 νησιά και βραχονισίδες. Από το σύνολο αυτών των νησιών κατοικούνται τώρα 115, το 2002 ήταν 127, δηλαδή παρατηρείται μια ερημοποίηση των νησιών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί άραγε. Παίρνουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες των νησιών που είναι αποκλεισμένα από τη θάλασσα. Ένα κοντέινερ για να έρθει από την Κίνα στον Πειραιά, το λιμάνι της Ελλάδος, το κεντρικό λιμάνι της Ελλάδος, κοστίζει 500 ευρώ. Για να πάει από το λιμάνι του Πειραιά σε ένα νησάκι που είναι γύρω στα 100 μίλια, κοστίζει 1500 ευρώ. Αυτό συμβάλλει στην ε, συνοχή. Ναι, τελειώνω κυρία Πρόεδρε. Ε, παράδειγμα, η, το καμποτάζ ε, το 2004 που ε, καταργήσαμε και εφαρμόζεται στην ε, χώρα μας αντί να έχει τα αποτελέσματα του ανταγωνισμού για να αυξήσει τις, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της θαλάσσιας μεταφορές είχε το ανάποδο αποτέλεσμα. Δημιούργησε μονοπόλια ε, δεν τους συμφέρει τους ακτοπλώου να πηγαίνουν στα μικρά νησιά γιατί δεν έχουν κέρδος και χρειάζεται να περιβαίνει το ελληνικό κράτος με χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σαν παράδειγμα το ανέφερα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Σερβία, κύριε Νικολίκη, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Στα πλαίσια αυτής της συνεδριάσεως και πέρα από την παρουσίαση του, της συναδέλφου του Σερβικού Κοινοβουλίου θα ήθελα να πω και εγώ κάποια πράγματα ότι τα Δυτικά Βαλκάνια και η Σερβία αντιμετωπίζουν προκλήσεις και θα αντιμετωπίσουν ε, προκλήσεις όσον αφορά τις μεταφορικές υποδομές. Συμπεριλαμβάνεται και χρονική περίοδος μετά το 2020 για να ξα... χρειάζονται οικονομικά ε, μέσα για υποδομές. Χρειάζεται, χρειάζονται έργα για την επόμενη περίοδο που θα χρηματοδοτούνται από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μέσω ταμείων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από το μέσο για τη σύνθεση της Ευρώπης και από το επενδυτικό πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων και κάποιο ποσό από τα χρήματα του προπολογισμού της Σερβίας. Πέρα από τα εθνικά οικονομικά μοντέλα για την υλοποίηση των έργων, θα υπάρξει και άλλο πρόβλημα. Η υλοποίηση των συμπράξεων ιδιωτικού δημοσίου τομέα για την ε, ε, χρηματοδότηση υποδομών και σχετικών έργων, μαζί με την υλοποίηση περιφερειακών έργων υποδομών στα Δυτικά Βαλκάνια, που θα είναι ένας από τους κλάδους των μελλοντικών TNT, θα είναι η κοινή αίτηση για τη ε, Ευρωπαϊκή Ενώσεων με γειτονικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για να στηριχθούν διασυνοριακά έργα που έχουν και περιφερειακή σημασία. Η υλοποίηση της, των μέτρων διασυ... μεταρρύθμισης διασυνδεσιμότητας για πιο εύκολη υλοποίηση των προγραμμάτων υποδομών που έχουν προτεραιότητα θα είναι άλλο ένα επικείμενο πρόβλημα και πρόκληση. Αυτά ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κράμερ, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό, κύριε Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση. Πάντα από τις αποτυχίες μαθαίνουμε εδώ και 22 χρόνια ψηφίσαμε το τούνελ ε, του Γκοτάρ. Η Ελβετία τελείωσε τη σύραγγά τη. Αντίθετα, τίποτα δεν έγινε από Ιταλική ή Γερμανική πλευρά. Και τώρα η Ιταλία πρέπει να χρηματοδοτήσει τη γραμμή διαδρομή Λιών Τωρίνο και η Γερμανία να χρηματοδοτήσει ορινά ορεινά περάσματα. Πρέπει να σταματήσουμε να γελάμε. Μήπως θα έπρεπε την επόμενη φορά να σταματάμε ένα πρόγραμμα πριν να ξεκινήσουμε 25 επόμενες, τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να μάθουμε τα παθήματά μας. Αναφέρθηκε ότι τα συνοριακά τμήματα είναι πολύ σημαντικά. Αλλά τα 90 μικρά προγράμματα που καταστράφηκαν για τα μεγάλα προγράμματα δεν συνεχίστηκαν. Ε, ε, ξεκινάμε, αφήνουμε μη τελεί κάποια προγράμματα που ξεκινήσαν πριν 30-40 χρόνια. Τα παρατάμε χωρίς να υπάρχει συνέπεια για την κινηματικότητα. Κινητικότητα, συγγνώμη. Θα πρέπει λοιπόν στην πράξη να βλέπουμε τι κάνουμε θα πρέπει να προστατεύσουμε την Ευρώπη και να εξασφαλίσουμε την κινητικότητα. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα ίδια σφάλματα του παρελθόντος, να μαθαίνουμε από τα παθήματα. Πρέπει να δράσουμε με ευφυΐα και σύνεση και να εφαρμόζουμε μικρά προγράμματα. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Ο κύριος Κώστα Σίλβα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους αγαπητούς συναδέλφους Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Ποια είναι η πιθανότητα όλα τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες πραγματικά να μπορούν να προχωρήσουν ταυτόχρονα ή μη, αν απλώς ε, ακολουθούμε προσέγγιση ανταγωνιστική, που πολύ συχνά συμβαίνει στην Ευρώπη, τότε θα χάσουμε την ευκαιρία για ε, να καλύψουν ανάγκες τους οι πιο αδύναμες περιοχές, οι πιο απομακρυσμένες περιοχές. Πραγματικά, να μπορέσουν να κινηθούν με την ίδια ταχύτητα όπως και πιο προοδευμένες περιοχές. Ε, τεχνολογικές υποδομές, πολυτροπικές ε, υποδομές, θαλάσσιες μεταφορές, σιδηρόδρομοι, περιβαλλοντικές πτυχές. Αν όλα αυτά είναι θετικά, το να δίνουν περισσότερα χρήματα είναι πολύ θετικό, αλλά συνοχή πρέπει να είναι το σύνθημα. Κινητικότητα, επίσης, Αλλιώς θα κινδυνεύουμε να αυξήσουμε τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών, ε, μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ ταχυτήτων των περιφερειών και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Λοιπόν, σας καλώ να εξετάσετε τα μέτρα, τα προγράμματα που αφορούν τις μεταφορές με έναν τρόπο συνεκτικό, να μην μένει κανείς πίσω. Ο κ. Στομά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε εδώ σήμερα το απόγευμα. Είναι εξέπαινη αυτή η πρωτοβουλία σας, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που την διοργανώσατε αυτή η συζήτηση. Συνάδελφοι, μιλάμε για τις υποδομές μετά το 2020. Και για να είμαστε επικοδομητικοί θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη σημερινή πραγματικότητα και την εξέλιξη των υποδομών μεταξύ Ανατολική και Δυτικής Ευρώπης. Πρέπει να ξέρουμε ότι η στρατηγική της Ευρώπης για μετά το 2020 για να επιταχύνουμε ακριβώς την ολοκλήρωση των υποδομών μεταξύ Ανατολική και Δυτικής Ευρώπης θα πρέπει να βασιστεί σε τρεις πυλώνες. Καταρχάς θα πρέπει να ε, ενθαρρύνουμε την διαδικασία προσχώρησης υποψηφίων χωρών, Ουκρανία, Μολδαβία κλπ. Στο πλαίσιο ακριβώς όπου θα έχουμε μια Ευρωασιατική Ένωση. Δεύτερον, θα πρέπει να εντάξουμε πλήρω τη χώρα Ανατολική Ευρώπη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει επίση να επιταχύνουμε αυτή την ένωση Ανατολική Δυτική Ευρώπη ώστε να υπάρχει μια αγορά και για τα εμπορεύματα αλλά και για τι επενδύσει. Και καταλήγοντα, κύριε Λολέια, θα ήθελα να σα ζητήσω, λαμβάνοντα υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, να συνοψίσετε τη στρατηγική για μετά το 2020 όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών για την Ανατολική Ευρώπη, λαμβάνοντα υπόψη ακριβώ τι υποψήφιε χώρε και τι χώρε τη Βορειοανατολική Ευρώπη. Ε, Ρουμανία, Μολδαβία, χώρε οι οποίε είναι ε, πολύ κοντά στι υποψήφιε χώρε. Για τον κύριο από την Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων, έχω μια ερώτηση. Η τραπέζα που εκπροσωπείται μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα που θα αφορούν αυτοκινητοδρόμους στην Ρουμανία με ΣΔΙΤ, με τη χρήση ΣΔΙΤ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιν Κάμπ. 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ τα Εθνικά Κοινοβούλια σήμερα, λέει ο κύριος Βαντερκάμπ. Πολύ καλό που έχουμε τη συζήτηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί σας. Δύο ερωτήσεις έχω στον κύριο Λελέη και μία στον εκπρόσωπό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πρώτη ερώτηση στον κύριο Γολολή. Είναι μια παρατήρηση πιο πολύ για το γεγονός ότι 60% του ΣΕΦ στο μέλλον θα πρέπει να δοθεί για την κλιματική αλλαγή και τις μεταφορές. Εσείς τι ακριβώς εννοείτε με αυτό. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε περισσότερο. Έπειτα, δεύτερη ερώτηση για σας. Δεν θα έπρεπε να δούμε όχι μόνο το θέμα των ε, επιχορηγήσεων, των ε, επιδοτήσεων. Νομίζω ότι σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο με αυτό και πολύ λιγότερο με τη λογική της δανειοδότησης. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είπε ο υπεύθυνο από το λιμάνι του Ρότερνταμ ότι οι εμπορικές τράπεζες συχνά ε, δεν βοηθούν αρκετά. Εσείς τι έχετε να σχολιάσετε για αυτή την παρατήρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βαντεγκάμ. Ο κύριος Ζωφ, εκεί είσαστε. Μάλιστα. Ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξότιμοι ευρωβουλευτέ, υπάρχει μια αντίφαση που ακούμε στι πολιτικέ επιλογέ όταν πρόκειται για τι υποδομέ μεταφορών. Γιατί από τη μια μιλάμε για επενδύσει για τον εξυγχρονισμό των υποδομών και των συστημάτων και από την άλλη έχουμε συγκεκριμένε εμπειρίε στην Πορτογαλία όλα αυτά τα χρόνια. Όμως έχουν μπλοκαριστεί οι επενδύσει. έχουν μπει όρια. Τα στοιχεία της Eurostat πριν από δύο μήνες έδειξαν ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν περισσότερα χιλιόμετρα στου από ότι ο δρόμους ε, χερσαίους, εκτός από την Πορτογαλία. Από το 2012 και μετά, λοιπόν, δημιουργήθηκε μια διάλυση του δημοσίου τομέα με την κρίση, δεν μπορούμε να προσλάβουμε υπαλλήλους κτλ. Οι πόροι κρατικοί εκταμιεύονται με το σταγονόμετρο. Υπάρχουν όρια στην Πορτογαλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα εκταμείευσης και χρήσης κονδυλίων για τέτοια προγράμματα υποδομών στις μεταφορές. Συνεπώς, μετά το 2020, τι θα γίνει. Θα πρέπει να δούμε ότι θα καταλήξουμε σε ασυμμετρίες. Ποτέ τα δημότικα ταμεία δεν μπόρεσαν να, να αντισταθμίσουν την διάλυση της χώρας, αλλά αυτά που προβλέπουμε για το μέλλον θα είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριος Μπάλσης. Λιθουανία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Όλουλα, κυρίω σε εσά απευθύνομαι. Μπορούμε να μιλούμε εδώ ώρες και ώρες και να λέμε τι ωραία που είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αν όμως δεν υπάρχουν χρήματα για τα προγράμματα αυτά, τότε είναι καταδικασμένα σε θάνατο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θέλω να πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΣΕΦ και την ε, συνοχή μετά το 2020 δεν φτάνουν και δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες της Λιθουανίας και άλλων χωρών συνοχής. 70% δεν φτάνει. Επιμένουμε λοιπόν να μείνει στο επίπεδο του 85% ώστε να υλοποιηθούν επιτυχώς τα προγράμματα αυτά. Έπειτα το σχέδιο για το Rail Baltic που θα συνδέει τις πρωτεύουσες τριών βαλτικών χωρών ε, με τη Φιλανδία και την Πολωνία. Όλος παραδόξως συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότης 85% μόνο ε, τα Λίν και Ρίγα, αλλά όχι αρνείται να χρηματοδοτήσει τη σύνδεση με τις άλλες πρωτεύουσε. Εκεί λέει στην καλύτερη περίπτωση 70%. Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και πρέπει να πω ότι εάν το ΣΕΦ δεν αναγνωρίζει τη σύνδεση με το Vilnius, ότι αποτελεί μέρος δηλαδή όλου του προγράμματος, τότε τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρο το Rail Baltica. Τι έχει να πει ο κύριος Ολέλε γι' αυτό. Έπειτα, η στρατιωτική κινητικότητα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας και θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον να χρηματοδοτηθεί. Όμως η συγχρηματοδότηση μέχρι 50% δεν φτάνει για τις χώρες συνοχές. Το ελάχιστο θα έπρεπε να είναι ή 70% που είναι ο μέσο όρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι Βαλτικέ χώρε είναι πραγματικά σημαντικέ για την Ευρώπη. Αν ναι, πρέπει να του δώσετε περισσότερη σημασία και να διατηρηθεί η έννοια τη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φίσρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα αρχίσω με το θέμα Λιόν Τωρίνο. Δεν πρόκειται για γαλλο-ιταλικό σχέδιο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Λιόν Τωρίνο είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και οικονομικά για τις συναλλαγές βορρά-νότου Ανατολής Δύσης, αλλά και περιβαλλοντικά. Υπενθυμίζω ότι η ρήπανση δεν γνωρίζει σύνορα. Σας καλώ να πάτε στη κοιλάδα Τόλπα για μια εβδομάδα και θα δείτε, θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο σχέδιο. Γι' αυτό και υπενθυμίσαμε στη Γερουσία, ο υπουργό δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι να γίνει το τούνελ αυτό και ότι έχει διεθνή διάσταση. Οι εργασίες θα πρέπει να προχωρήσουν το 2018. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση, αυτό είναι κάτι γαλλογαλλικό όντως. Εμείς θελήσαμε να αναβάλουμε κατά κάποιο τρόπο την πρόσβαση για να προσαρμοστούμε στον καινούριο αριθμό των τρένων, γιατί η υποδομή μέχρι τώρα δεν ανταποκρίνεται. Τώρα η εκτίμηση που έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. έχει αναγνωρίσει τις επιτυχίες ε, των ε, επενδύσεων. Οπότε στηρίζω τη βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει σχέδια με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, αλλά και σχέδια που οδηγούν τις μεταφορές εκτός ε, οδικών δικτύων. Είναι πολύ σημαντική και η χρηματοδότηση για τον εξυγχρονισμό αλλά λυπάμαι που βλέπω ότι δεν υπάρχει αρκετή φιλοδοξία στην οικονομική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τα κονδύλια. Τέλος, για την υλοποίηση πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να υπάρχει μεγαλύτερη προβολή και όπως πρόσφατα ακούσαμε ότι πρέπει να μπορούμε να κυκλοφορούμε στην Ευρώπη και να τη διανύουμε χωρίς να την καταστρέφουμε. Ο κύριος Σανστέρ, πού είναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω και εγώ δύο λόγια παρά αυτά που ο άλφος από τη Λιθουανία σε σχέση με την χρηματοδότηση και το νέο πι για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας λοιπόν είναι απαραίτητα τα κονδύλια αυτά ώστε να φέρουμε πιο κοντά τους Ευρωπαίους και να επικεντρωθούμε ακριβώς στην προσθέμενη αξία των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Έχουμε ευκαιρίες επενδύσεων σε αυτά τα διασυνοριακά προγράμματα, οπότε θα ήταν καλό η Ένωση να στηρίξει την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Η διευκόλυνση του συνδέοντα στην Ευρώπη ήταν χρήσιμη για την εφαρμογή προγραμμάτων που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη. Οπότε χαίρομαι που η Κομισιόν πρότεινε να συνεχιστεί το ΣΕΦ, το πράγμα ΣΕΦ, στο επόμενο ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ Με σημαντικό βαθμό συγχρηματοδότησης, δημιουργώντας έτσι την βάση για την επένδυση σε υποδομές σε χώρες συνοχής νέα στοιχεία όπως η κατανομία ανα βαθμό ανταγωνιστικότητα, η στρατηγική κινητικότητα, κινητικότητα και άλλα στοιχεία είναι ευπρόσδεκτα. Είναι επίση σημαντικό προγράμματα τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του τωρινού πι να ολοκληρωθούν στα πλαίσια του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα διέρχεται λοιπόν το δίκτυο αυτό από όλες τις χώρες της Βαλτικής και θα περιλαμβάνει και την Πολωνία και την Φιλανδία δημιουργώντας ένα σοβαρό οικονομικό διάδρομο. Η προσθέμενη λοιπόν αξία είναι προφανής και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Merci beaucoup et je inscrite. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ έβαλα τον εαυτό μου στον κατάλογο των μιλητών και επίσκο συμφωνώ η συζήτηση είναι μόνο για το Λιόν αλλά εδώ έχουμε μια προβληματική που αφορά όλες τις χώρες, δηλαδή την ρήπανση. Εκτός και αν θέλουμε να περιμένουμε το 2026 για να ασχοληθούμε με τη ρήπανση. Μέχρι τότε όμως τι κάνουμε δεν είναι να μην συζητάμε καθόλου για αυτό το θέμα. Η τερύπανση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε άμεσα, γιατί είναι θέμα δημόσια υγεία και νομίζω γι' αυτό συμφωνούμε όλοι. Να σα πω λοιπόν, κύριε, ότι σήμερα χρειαζόμαστε κάποια αποτελεσματικότητα. Το είπατε και εσείς. Κάτι που μας επιτρέπει βεβαίω να ενισχύσουμε το δίκτυο και την σύνδεση, τη διασυνοριακή. Όμως, όμως, βεβαίως, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα ευρωπαϊκά εργαλεία με τρόπο αποτελεσματικό, αλλά να μην ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε τα διορθωτικά ταμεία επενδύσεων, ταμείου συνοχής, ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία και για τις δικές σας περιοχές έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κινητικότητα. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, εγώ πιστεύω πολύ στην συνδυασμένη προσέγγιση διαφορών χρηματοοικονομικών εργαλείων το blending όπως το λέμε. Προσοχή όμως, το blending αυτό, αυτός ο συνδυασμό να μην παραβλέπει το ότι καταρχάς χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό προπολογισμό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αν πούμε ότι μην στεναχωριέστε, θα κάνουμε του κατάλληλου συνδυασμού κτλ. χωρί να το πηγαίνετε σε προπολογισμό, διαφωνώ. Γιατί διαφωνώ. Γιατί απλούστατα κατά τη διάρκεια τη τρέχουσα περίοδου, εμεί παραχωρήσαμε ένα σημαντικό κομμάτι του μηχανισμού διασυνδεσιμότητα για να πάμε στο σχέδιο που ονομάσαμε σχέδιο Juncker, στο ΕΦΣΥ. Αν εσεί λοιπόν δείτε τώρα το ΕΦΣΥ, το σχέδιο Juncker, και δείτε ας πούμε το ποσοστό που πάει στα προγράμματα μεταφορών, στα έργα μεταφορών είναι 9% μόνο. Ε, δεν γίνεται. Εγώ θα ήθελα στον επόμενο προγραμματισμό να πάμε όχι μόνο στο 9% για τις μεταφορές, να πάμε τουλάχιστον σε ένα 20, 30 και 40 μάλιστα για τα προγράμματα μεταφορών. Και τέλος, καταλήγω, όχι δεν καταλήγω, τα πάω όλα γιατί καθυστέρησα. Λοιπόν, κύριοι, είχατε πολλές ερωτήσεις και δεν έχετε παρά δύο λεπτά για να απαντήσετε ο καθένα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Κύριε Λάι, έχετε εσεί πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σα ευχαριστήσω για τις πολλές ερωτήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται τουλάχιστον μισάωρο. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να τα απαντήσω όλα αυτά στα δύο λεπτά. Παρ' όλα αυτά σημαντικά, σημαντικά πράγματα υπόθηκαν. Συνέργειε, βεβαίω, βεβαίω. Το τόνισα και εγώ. Είπα ότι όταν μιλάμε για προγράμματα μεταφορών θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα τη σφαιρική, τη γενική εικόνα, the big picture, ε, ψηφιακή υποδομή των προγραμμάτων κλπ. Όταν μιλάμε για την αποανθρακοποίηση, αποανθρακοποίηση και ψηφιοποίηση είναι τα δύο κύρια στοιχεία τη πολιτική τη Ένωση για τι μεταφορέ. Το οποίο σημαίνει ότι η χρηματική το οικονομική υποδομή θα πρέπει να στηρίζει αυτές τις δύο πτυχές. Άκουσα προηγουμένως για το μέχρι 60% ας πούμε περιβαλλοντικής στήριξης. Δεν είναι ότι ξαφνικά γίναμε όλοι οικολόγοι, καλό θα ήταν βέβαια, αλλά σημαίνει ότι εμείς στηρίζουμε αυτό το είδος προγραμμάτων υποδομής που έχουν μέγιστη απόδοση και επιδόση όσον αφορά την αποανθρακοποίηση του τομέα των μεταφορών που έχει υψηλέ εκπομπές διεξιδίου άνθρακας, το οποίο σημαίνει ότι στηρίζουμε ας τον συνδρόμο και οποιαδήποτε άλλη μορφή καθαρής μεταφοράς, καθαρών μεταφορών. Το ίδιο για τις συνέργειες. Κάνουμε το ίδιο για τα αναλλακτικά καύσιμα, ας πούμε. Γιατί στηρίζουμε την υποδομή για τα αναλλακτικά καύσιμα, για, την, για το λεκτικό ρεύμα, για το φυσικό αέριο κλπ. Ταυτόχρονα όμως, συνδυάζοντα στηρίζουμε και την ψηφιοποίηση. Γιατί όλα αυτά είναι νέα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με παλιού τρόπου, με παλιέ νοοτροπίε. Πρέπει να βρούμε νέε νοοτροπίε. Αυτά πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε, γιατί να συνδυάσουμε όλα αυτά, Συνέργειε από ανθρακοποίηση κλπ. Επίσης, με τα διάφορα άλλα εργαλεία. Εργαλεία τα οποία μπορούν να μας ωφελήσουν. Το συνδέω στην Ευρώπη, ε, ο Ορίζοντας, ε, το Ταμείο Συνοχής, ε, το ΕΦΣΙ, όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν. Και συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε στο ΕΦΣΙ περισσότερα προγράμματα για τις μεταφορές. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το ρυθμό μας οι επιδοτήσει δεν, ε, παλιά μάλλον ήταν συνώνυμο των μεταφορών, Όμω έχουν αλλάξει οι καιροί. Πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί. Θα πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί και στο blending, στο συνδυασμό, θα πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί στο να εμπλέξουμε τον ιδιωτικό τομέα και τις επενδυτικέ τράπεζες. Μεγάλη αλλαγή λοιπόν και αυτή. Και επίση τότε μόνο θα μπορούσαμε να πάμε σε αυτά τα επίπεδα και να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση. Και σας παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι έχουμε λιγότερα χρήματα στον προπολισμό από ό,τι είχαμε στον παρελθόν και έκανε καλή δουλειά η Κομισιόν που κατέθεσε μια πρόταση η οποία είναι βαρύς. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια πρόταση η οποία χρειάζεται αλληλεγγύη, όχι μόνο αλληλεγγύη σε σχέση με τους ωφελούμενους, αλλά και σε σχέση με τους δωρητές. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια διαβάθμιση. Δεν συμφωνώ ότι υπάρχουν λιγότερα για τις μεταφορές, 20% μάλλον παραπάνω από ό,τι είχαμε στον προηγούμενο προπολογισμό. Αυτή είναι η πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δηλαδή έχουμε κάτι το οποίο το έχουμε τεντώσει. Και όλος ο προπολογισμό της Ένωσης έχει διαφορές είναι τελείως διαφορετικός όσον αφορά ταμεία, συνοχής, ε, τις χρηματοδότητες κτλ. Δεν έχουμε τα ίδια ποσοστά ε, συγχρηματοδότηση από ό,τι έχουμε στο Ταμείο Συνοχής. Ταυτόχρονα όμως κάνουμε πιο έντονους τους δεσμούς, τους ενοριακούς. Γιατί άκουσα από τον Δανό συνάδελφο προηγουμένως που έλεγε ότι αυτοί έχουν μεγάλη προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Οπότε, συνοχή, 85%. Ε, το ίδιο στα δύο ε, ποσοστά τα οποία χρηματοδοτούνται από το Γενικό Ταμείο ΣΕΦ. Θα έπρεπε λοιπόν να επικεντρωθούμε περισσότερο και να αντίνουμε το διασυνοριακό στοιχείο. Και άκουσα από τον Λιθουανό συνάδελφο αυτά που είπε για τη Βαλτική και το πρόγραμμα που είναι ανταγωνιστικό και περιλαμβάνει πέντε χώρες και έχει πολλές καλές πιθανότητες να συνεχίζει να χρηματοδοτείται από την επόμενη διαυκόλυνση του προγράμματος συνδέοντας την Ευρώπη. Πρέπει επίσης να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό, το έργο αυτό, να προχωρήσει ώστε να έχουμε επιτέλους αυτό τον άξονα βορρά-νότο. Για το Βίλνιους, ας πούμε, αν δούμε τη χρήση των χρημάτων των Ευρωπαίων θα πρέπει να αναζητήσουμε την βέλτιστη οδό χρηματοδότησης. Και βεβαίως του του υπάρχουν και άλλοι τρόποι χρηματο... Ε, χρήση αυτών των υπόλοιπων χρηματοδοτικών εργαλείων. Πρέπει να τα συνδυάσουμε απλά και μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Το συντρίψατε το, το σκορ του χρόνου αγόρευσης. Κύριε Σίμψον, έχετε το λόγο. Και μετά θα κλείσουμε τον επόμενο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν πολλέ ερωτήσεις που μου απευθύνθηκαν. Άρα όλοι υποστηρίζουν τους αυτοκινητόδρομους τη θάλασσα, έτσι το εκλαμβάνω. Αλλά προσβλέπω σε μεγάλη ζωή χρημάτων και πολλά πολλά ακόμα έργα και, προγράμματα. Κάτι είπε ο Έλληνα συνάδελφος που είναι πολύ σημαντικό. Οι περιφερειακέ οι απόμακρες περιοχέ, Διότι οι περιφερειακέ περιοχέ δεν συμπεριλαμβάνονται στους βασικούς κεντρικούς χάρτες. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα με μένα και για την βραχή αναψυπλοεία. Και με το πρόγραμμα εφαρμογής μου συγκεκριμένα αναφέρω τις περιφερειακές περιοχές, τα νησιά της Ελλάδας και τα νησιά της Ισπανίας, Κανάρια κλπ. Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ιμπίθα στην Ισπανία. Και με το Brexit το νησί της Ιρλανδίας γίνεται περιφερειακή περιοχή. Άρα πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους πώς αυτές τις περιοχές θα τις εντάξουμε στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, το TNT. Ο συνάδελφος από τη Φιλανδία, στο τελευταίο πάνελ, είπε, αναφέρθηκε στη Φιλανδία και την παγωμένη Βαλτική και δώσαμε επίσης τα παγωθαυστικά χρήματα εκεί, από τους αυτοκινητόδρομους της θάλασσας. Εγώ προσπάθησα να πείσω τον Κύπριο, είχα πρόβλημα να πείσω τον Κύπριο Υπουργό Μεταφορών, χρειαζόμαστε παγωθαστικά, πού να τον πείσω, τελικά τα κατάφερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να παραμείνει ανοιχτή η ναυσιπλοεία στη Βαλτική. Πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά την ναυσιπλοεία στα βόρεια της Ευρώπης είσαστε από κοινοβούλια των κρατών μελών. Θα με συγχωρήσουν οι πρώην Ευρωβουλευτέ. Εσεί από τα κράτη-μέλη, από τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Ό,τι αποφασίζετε, αποφασίζετε από την κυβέρνησή σα, από τι κυβερνήσει σα. Εσεί έχετε ρόλο να παίξετε, να πιέζετε τι κυβερνήσει σα για αυτό που θέλετε και για να πιέσετε τι κυβερνήσει σα για περισσότερα χρήματα για, τις αυτο... για και να πούν στο Χένρικ θέλουμε περισσότερα χρήματα για αυτοκινητόδρομου τη θάλασσα. Λοιπόν αυτό θέλουμε, ας τα πάρουμε. Καλό να πηγαίνει κανείς στις ε, αυτέ εκδηλώσει και να λέει αυτό που λέει και όταν επιστρέφετε να πηγαίνει στις πατρίδε σα. και να μην στηρίζετε τα λόγια σας, αυτά που λέτε εδώ, δεν τα υλοποιείτε. Στηρίξτε παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις μάχες που δίνει με το Συμβούλιο για τον προπολογισμό και σας παρακαλώ, σας εκλυπαρώ, πηγαίνετε στις κυβερνήσεις σας και στηρίξετε πρώτα τους αυτοκινητόδρομους της θάλασσας, αλλά όλους τους διαδρόμους να στηρίξετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σίμψον. Λοιπόν, όταν λέτε, σα λένε υποστηρίξτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υποστηρίξετε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι διαπραγματεύσει μετα... γίνονται μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, έτσι. Συμφωνούμε, έτσι, κύριε Σίμψον. Ναι, ναι, συμφωνούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κύριε Ντάνετ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ να απαντήσω σύντομα στις ερωτήσεις σας. Στον κύριο Κράμερ, μικρά προγράμματα. Ναι, ενδιαφέρεται για μικρά προγράμματα η τράπεζα. Έχουμε προϊόντα τα οποία συσσωρεύουν μικρά προγράμματα, τα κάνουμε καλύτερα και αυτό έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά πολλές φορές. Ε, ο κύριο Στόμα, Ρουμανία, για τη χρηματοδότηση. Όταν παίρνουμε ένα αίτημα για χρηματοδότηση, το εξετάζουμε σύμφωνα με τα συνηθισμένα μας τεχνικά κριτήρια δανεισμού. Πάντως, κύριε Βαντεκάμ, για το θέμα των επιτοκίων. Δεν θέτουμε επιτόκια εμείς, δανειζόμαστε από τις αγορές. Αυτό είναι το κόστος του δανεισμού. Το business ε, model μας είναι το τριπλό α, οπότε μπορούμε να δανειστούμε φτηνά, όπως κάθε τριπλό α. Και μετά τα δίνουμε τα χρήματα ως δημόσιος που είμαστε στους δανειζόμενους. Δεν είναι τόσο το θέμα των επιτοκίων, όσο είναι ε, οι συνθήκες δανεισμού που είναι μακροχρόνιες. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, για το σχέδιο Juncker, στόχος ήταν να δοθούν κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις στην οικονομία. Εξαιτία της δομής των μεταφορών, πολλές επενδύσεις γίνονται από το δημόσιο τομέα. Αν θέλουμε μεγαλύτερο κομμάτι ε, μηχανισμών ε, Ταμείου Juncker, ε, τότε θα πρέπει να αλλάξει και η λογική της χρηματοδότησης. Ευχαριστούμε. Ωραία. Μπορούμε να τους χειροκροτήσουμε τον κύριο Χολέλα, τον κύριο Σίμψον και τον κύριο Ντάνετ. Ε, ευχαριστούμε πολύ που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, έτσι. Θα έχουμε την ευκαιρία πάλι. Η συζήτηση αυτή για τον προπολογισμό μόλις αρχίζει όπως καταλαβαίνετε και τώρα περιμένουμε, όλοι τον περιμένουμε τον κύριο Είναι εδώ. Ωραία. Thank you. you Monsieur Tinger, bonsoir. Κύριε Τιγκέρ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας προσκαλέσαμε για ερωτήσεις, απαντήσεις με τον Επίτροπο δηλαδή που είναι υπεύθυνο για τον προπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή μου, η Επιτροπή Μεταφορών, ξέρετε ότι είναι αποφασισμένη να φροντίσει να υπάρχουν κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό να έχουμε πρόγραμμα, μηχανισμούς διασύνδεσης που να είναι σύγχρονοι, που να τα αποκρίνονται στις ανάγκες. Δεδομένου μάλιστα ότι για όλους είναι απαραίτητο να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης να ολοκληρωθούν τα δίκτυα και υποδομές στις περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης. Να μην ξεχνάμε ούτε τις, τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας, αλλά ούτε και το σύστημα διαχείρισης των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Δεν έχουμε μιλήσει, με το... Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τους ενιαίους εθέρες και την ψηφιακή διαχείριση Οπότε κύριε Τιγκέρ, περιμένουμε ανυπόμονα να σας ακούσουμε, να μας πείτε εσείς πώς βλέπετε τις μεταφορές, ώστε να προχωρήσουμε στο θέμα των ευρωπαϊκών υποδομών και ποια θα είναι ακριβώ τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα στηρίξουν μετά το 2020. Γιατί για τον προπολογισμό τα πράγματα είναι δύσκολα. Ε. Λοιπόν, 10 λεπτά κύριε Τιγκέρ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια επίσης. Καλησπέρα. Η σημερινή σας συνάντηση έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή που αρχίζουμε να συζητάμε για το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη δεκαετία. Η Ευρώπη ήταν και παραμένει η ήπειρος του μέλλοντος. Μετά την ε, γερμανική ήττα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ανάμεσα στο Κέλ και το Στρασβούργο, διακόπτηκε η σύνδεση παντελώς. Οι γέφυρες καταστράφηκαν, έπεσαν. Μετά είχαμε τον ψυχρό πόλεμο, και με το Στάλιν δεν υπήρχε καν λιμάνι στην περιοχή κοντά στη Γερμανία. Υπήρξε δηλαδή μεγάλο πρόβλημα έλλειψης διασύνδεσης. Οπότε πρέπει να ξαναχτίσουμε τις υποδομές, να ξαναφτιάξουμε γέφυρες, για τους σιδηροδρόμους, να υπάρχει πάλι σύνδεση με θαλάσσιες μεταφορές και να διασφαλίσουμε και την ψηφιακή συνεργασία. Στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό θέλουμε να προβλέψουμε προγράμματα όπου η Ευρώπη να αποτελεί πραγματικά την προστιθέμενη αξία. Προγράμματα δηλαδή όπου η Ευρώπη συντονίζει το σχεδιασμό, όπου η Ευρώπη θα είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα 28-27 χωρών μελών. Και βέβαια αυτό θα γίνει πολύ καλύτερα εφόσον υπάρχει συντονισμός. Η Ευρώπη είναι μια εσωτερική αγορά και υπάρχει ελεύθερη διακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων. Πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Εμείς ως ε, παραγωγή και ως και καταναλωτές αποτελούμε πλήρως μέρος της εσωτερικής αυτής αγοράς. Έχουμε ποτά, φρούτα, λαχανικά, ρούχα, τα οποία παράγονται παντού στην εσωτερική αγορά και καταναλώνονται και παντού, πουλούνται παντού. Πρέπει να βαθύνουμε περισσότερο λοιπόν στο θέμα του πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις μεταφορές. Πώς μπορούμε να περιορίσουμε την ε, μετακίνηση σε ένα τμήμα μιας πόλης, για παράδειγμα. Όμως ο άνθρωπος, ο πολίτης, θέλει να συνεχίζει να έχει την ελευθερία να κυκλοφορεί και να μετακινείται, να πηγαίνει όπου θέλει και να αγοράζει ό,τι επιθυμεί. Οπότε η ανάγκη υποδομών μεταφορών μπορεί με να μειωθεί, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να διατηρήσουμε και να επαναδιοργανώσουμε τις υποδομές μας. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα σιδηροδρόμων λοιπόν αποτελούν δίκτυα για τους πολίτες και για τα εμπορεύματα. Είναι μια ευφύης έννοια. Έχουμε το δίκτυο ΚΑΝ, το οποίο θέλουμε να διευρύνουμε 2020-2030, με στόχο να ολοκληρωθούν ε, τα δίκτυα μέχρι το 2050. Στην ε, διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη έχουμε κάνει προτάσεις για την ανάπτυξη των δικτύων τα επόμενα χρόνια. Έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα από τις εμπειρίες που είχαμε μέχρι τώρα για τη συγχρηματοδότηση, το συνδυασμό χρηματοδότησης καθίσαμε και σκεφτήκαμε τι έχει γίνει και από πλευρά συντονισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε στρατηγικό πρόγραμμα έχει ένα συντονισμό. Οι περιφέρειες, οι χώρες μέλη πρέπει να στηρίζουν τα προγράμματα αυτά με ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Πριν από 20 χρόνια και ακόμα παραπάνω είχαμε μιλήσει για το, τη βιομηχανική σύνδεση από το Ρότερνταμ, Άμστερνταμ, Ρίνο... Ε, διασυνδέσεις που περνούσαν από τις Άλπεις. Όμως, δυστυχώς, δεν δόθηκαν όλες οι άδειες. Οπότε από τα μεγάλα αυτά σχέδια που είχαν προβλεφθεί, τελικά μόνο το τούνελ κοντά έγινε. Και το έκαναν οι Ελβετοί. Κρίμα δεν είναι. Η Ιταλία, η Γερμανία δεν προχώρησαν πολύ στα μεγάλα αυτά σχέδια και προγράμματα. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει καλός συντονισμός στο σχεδιασμό. Καλός συντονισμός πρώτα απ' όλα στο πρώτο στάδιο αδειοδότησης. Γιατί από εκεί ξεκινάει η δημιουργία των υποδομών. Ο συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι κέριος. Πρέπει να προβλέψουμε επίση και ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. Γι' αυτό εμείς προβλέψαμε ότι το ΜΕ e παρά το Brexit δεν θα περιοριστεί διότι θα έχει έναν ικανοποιητικό προϋπολογισμό για τους σιδηροδρόμους, για τις οδικές μεταφορές, για την ενέργεια και για τα ψηφιακά. Έχω μιλήσει πολύ με τις διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θέλουν να αναπτύξουν διασυνοριακές υποδομές. Για παράδειγμα, το Rail Baltica ανάμεσα στη Φιλανδία και την Εστονία τη Λετωνία, Λιθουανία και Πολωνία. Εδώ πρόκειται για ένα σχέδιο που δεν υπάρχει ακόμα ικανοποιητική υποδομή. Προβλέπεται ένα σχέδιο αγωγών προκειμένου να μην υπάρχει εξάρτηση αποκλειστικά και μόνο από τη Ρωσία της περιοχής αυτής. Πολύ σημαντικό αυτό. Η σύνδεση με τη Βόρεια Γερμανία και Δανία είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ε, το τούνελ στην Ιταλία επίσης είναι πολύ σημαντικό. Συνεπώς, έχουμε διάφορα σχέδια, τα γνωρίζουμε, ε, τα δέχτηκαν οι χώρες μέλη και τώρα πρέπει να προβλεφθεί ίση χρηματοδότηση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Όλα αυτά τα σχέδια αποτελούν προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. Πέρα λοιπόν από αυτό το ΕΜΑΗ, εμείς προτείνουμε τα προγράμματα συνοχής να υποφεληθούν από μεγαλύτερο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Μιλάμε βέβαια για 27 χώρες μέλη, έτσι. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές και οι οδικές μεταφορές είναι υπηρετικές, εννοείται. Κοιτάξτε, σκεφτόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει προσχώρηση της Μακεδονίας, Βοσνίας, Αγωβίνης, Κωσυφοπεδίου, Μαυροβουνίου κτλ. Εφόσον γίνουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουν προηγηθεί υποδομές. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν πρέπει να εμποδίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία. Και το θέμα της συνεργασίας Αυστρίας, Σλοβενίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Ελλάδας και των υποψηφίων χωρών είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει. Θέλουμε να προβλέψουμε το καμποτάζ να αναπτύξουμε καλά ενεργειακά δίκτυα. Και επίσης πρέπει να φροντίσουμε οι ροές μεταφορών να γίνονται όσο γίνεται καλύτερα. Να είναι ψηφιακή η διαχείριση της κυκλοφορίας. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και την λειτουργία των αυτόνομων οχημάτων, ε, της ε, συμπόρευσης, σύμπλευσης πολλών μέσα στο ίδιο όχημα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Τα δίκτυα επικοινωνίας της πέμπτης γενιάς είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε 27 διαφορετικές προσεγγίσεις στην Ευρώπη. Όχι. Τελεία. Ο συντονισμός πρέπει να γίνεται σε επίπεδο υπήρου και Ευρώπης. Ακόμα και η Ρωσική Ομοσπονδία συμπεριλαμβάνει την Ουκρανία και παρά τις κυρώσεις υπάρχουν εκατοντάδες φορτηγά τα οποία καθημερινά κυκλοφορούν από την Αγία Πετρούπολη ε, στην ε, Πολωνία, στο Κίεβο κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να συνδυαστεί και το πρόγραμμα αυτό με το Invest EU. Έτσι, με αυτή την προσέγγιση πρέπει να προχωρήσουμε. Και ολοκληρώνοντας, η εξέλιξη των υποδομών στην Ευρώπη και προς την Ευρώπη δεν πρέπει να μείνει στα χέρια μόνο των Κινέζων. Υπάρχει ο δρόμος του μεταξιού. Δεν πρέπει όμως να πουλήσουμε τη στρατηγική μας. Ούτε να αφήσουμε τους δρόμους μας και τις διαδρομές μας σε μη Ευρωπαίους. Πρέπει να παρεύουμε, πρέπει να εξασφαλίσουμε την κυριαρχία μας στον τομέα της κινητικότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ψηφιστεί ότι θα μείνουν τα δίκτυα αυτά σε ευρωπαϊκά χέρια. Διότι η Ευρώπη δεν θέλει να εξαρτάται από άλλους. Θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Και τέλος, το τελευταίο. Για τη Βία Μπάλτικα. Εάν θέλουμε να περάσουμε από το στάδιο του σχεδιασμού στο στάδιο της, ε, των προσφορών, δεν πρέπει να περιμένουμε άλλα 10 χρόνια. Όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, τόσο το καλύτερο. Γι' αυτό ε, σα ζητώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξετε το δικό μου φιλόδοξο σχέδιο ΣΕΦ για τον προϋπολογισμό από το 2021 και να εγκρίνεται το σχέδιό μου πριν από τις εκλογές του 2019. Γιατί αλλιώ πρέπει να περιμένουμε το Δεκέμβριο του 2020 για να γίνει κάτι. Και βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε η επόμενη πλειοψηφία που θα έρθει εδώ τι θα κάνει. Δεν ξέρουμε τι δυνατότητες χρηματοδότησης θα έχουμε αν καθυστερήσουμε και περιμένουμε. Η στρατηγική σημασία υποδομές είναι το καλύτερο παράδειγμα. Η έγκριση του ευρωπαϊκού προπολογισμού πρέπει να γίνει πριν από τις επόμενες εκλογές. Αν καθυστερούμε και αργήσουμε να εγκρίνουμε τον προπολογισμό, αυτό θα ήταν πάρα πολύ αρνητικό για την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και πολιτών. Και τέλος, για τη συζήτηση που γίνεται αυτή την εποχή. Πιστεύω ότι πρέπει να ελέγχουμε τα εξωτερικά μας σύνορα για να ξέρουμε ποιος έρχεται στις χώρες μας, ποιος μπαίνει. Και στα εσωτερικά σύνορα δεν πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, γιατί αν όλο και περισσότερο επανέλθουν τα εσωτερικά σύνορα σε εθνικό υπερφαριακό επίπεδο, τότε οι καλύτερες υποδομές μεταφορών θα είναι άχρηστες, γιατί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ε, συμφορήσεις, επειδή θα υπάρχουν έλεγχοι, τα προϊόντα θα μπλοκάρονται μέσα στα φορτηγά και οι πολίτες μέσα στα αυτοκίνητά τους. Στη Βαβαρία, στη Γερμανία και στην Αυστρία και αλλού έχει συζητηθεί πολύ το θέμα του ελέγχου των συνόρων και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν νέος που υπήρχε έλεγχο στη Βάδη στην ε, Γερμανία. Και τώρα, από τότε που υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία, ε, ανάμεσα στην Αλσατία και την Βαδιβλημέρ και τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και τα εμπορεύματα φτάνουν έγκαιρα στον προορισμό τους. Χρειάζεται όμως έλεγχος των συνόρων στο εξωτερικό, των εξωτερικών συνόρων. Αυτό είναι καλύτερο και είναι καλύτερο και για τις υποδομές. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Με τα σας ακούμε ότι ο προπολογισμό για το μηχανισμό διασύνθεσης δεν θα μειωθεί. Αλλά βέβαια υπάρχουν και ερωτήσεις. Θα σας θέσουμε τις ερωτήσεις κυρία Έντιγκερ. Να δώσουμε το λόγο σε εσά, τον κύριο Μπρέντ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την εδώ Ευχαριστώ λοιπόν τον Επίτροπο για την παρέμβασή του που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση, για τις φιλοδοξίες που εκφράσατε για το μέλλον. Εγώ σαν δανός με τα χαράς άκουσα που λέτε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή, ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τις υποδομές μας και να μην τις αφήσουμε τις υποδομές μας σε άλλους. Συμφωνούμε απόλυτα εδώ. Είναι Κάτι το οποίο συμφωνούμε πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες επί των ευρωπαϊκών υποδομών. Ήδη ακούσαμε στις συζητήσεις αυτά που είπε και ο Μπράιν Σίμψον, ότι οι χώρες θα πρέπει να παρέμβουν και αυτές, ότι έχουν ευθύνη. Έχω μία ερώτηση για ένα θέμα που δεν έχουμε συζητήσει ακόμα. Οι όροι για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να έχουμε και εμεί ήδη δική μα χρηματοδότηση. Με τη δημοσιονομική πειθαρχία που έχουμε όμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τι συμφωνίε που έχουν συναυτεί μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, με όλα αυτά κινδυνεύουμε να υπονομεύσουμε προγράμματα που θα έπρεπε να ενισχύσουν την κινητικότητά μα και θα έπρεπε να είναι καλά προγράμματα για το περιβάλλον και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν απασχόληση και θα μπορέσουν να καταπολεμήσουν τη συμφόρηση και θα μπορούσαν αυτά τα προγράμματα να μπλοκαριστούν και αυτό διότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε οικονομίες, ατέρμονες οικονομίες. Σαν επίτροπο, θα ήθελα να το σκεφτείτε καλά το θέμα τη χρηματοδότηση, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, ακριβώ ένα λεπτό. Ο κ. Μαρινέσκου, έχετε το λόγο για ένα λεπτό κι εσεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για τι προσπάθειέ σα Ξέρουμε ότι είστε σε πολύ δύσκολη θέση, προσπαθείτε να πείσετε όλα τα κράτη-μέλη να δώσουν περισσότερα χρήματα. Αλλά να λέτε ότι ο ΣΕΦ δέχτηκε γενναιόδωρο προπολογισμό, είναι υπερβολικό. Ε. Να σα υπενθυμίσω ότι το 2011 οι πρώτε ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν 50 δι σε σταθερές τιμές. 54. Τώρα είναι 42. Μετά από 7 χρόνια είναι λιγότερο το ποσό από ό,τι ήταν το 2011, διότι τότε ο Κάμερον μείωσε τον προϋπολογισμό και η μεγαλύτερη μείωση έγινε στον τομέα των μεταφορών. Τώρα είναι 42. Καλώς. Ε, δεν είναι αρκετά τα χρήματα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επενδυτικές ανάγκες που έχουν υποδομές. Έχω μία ερώτηση, συντομότατη. 6,5 δις. Αυτό είναι το τμήμα της αύξησης για στατιωτική κινητικότητα. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας στον κανονισμό. Περιμένετε από εμά να, να θεσπίσουμε τους κανόνες. Αλλιώς θα είναι μόνο για στατιωτικούς σκοπούς και όχι για το ΣΕΦ δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα. Εμείς θα προτείνουμε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα βέβαια. Δεύτερον, εν γέννη, σε όλους τους οριζόντιους κανονισμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πολλές εφαρμοστικές πράξεις, όχι κατά εξουσιοδότηση Και πολλά γενικά σχόλια στο διατακτικό του κανονισμού. Τι σημαίνει αυτό ότι θέλει να ηγηθεί όλων των προγραμμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι θέλει χωρίς το Κοινοβούλιο, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα να κλείσουν αυτά τα χαρτοφυλάκια πριν τις εκλογές, εάν ισχύει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Κύριε Καματερέ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, ε, για πείτε μου, τι προβλέπετε στον προϋπολογισμό ε, για την αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος. Ε, είπατε, από ό,τι κατάλαβα, για ενίσχυση της φύλαξης ε, στα σύνορα. Νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μάισνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καλή ομιλία ευρωπαϊκή, ήταν αυτή που κάνατε, αλλά έχω δύο ερωτήσει. Είπατε ότι δεν θα υπάρξει μείωση. Είσαστε σίγουροι ότι θα σα ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη, διότι καμιά φορά συμφωνούν το Ευρωκοινοβούλιο και, το και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μειώνουν τα κράτη-μέλη του προπολογισμού. Μετά είπατε ότι τα χρήματα θα πήγαιναν για δρόμου, για σιδηροδρομικέ ε, γραμμέ και για τι θαλάσσιε μεταφορέ. Στον αφορά του θαλάσσιου αυτοκινητόδρομου. Συγγνώμη, τέλο πάντων, του διαδρόμου αυτού του θαλάσσιου. Τι θα γίνει, πώ θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι. Ευχαριστώ κύριε Μάσινο. Κύριε Κράμερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο Έλβα ήταν στο ψυχρό πόλεμο το σύνορο και όχι το Ομπεράιζα. Αλλά τέλο πάντων, έχουμε αυτά τα διασυνοριακά προγράμματα και με κονδύλια ευρωπαϊκά έχουμε χρηματοδοτήσει μέχρι το Κατόβιτσε δημιουργία σιδηροτροχιών, Αμβούργο, Κρακοβία, ε, συνεχόμενη εξέλιξη του σιδηροδρόμου. Πέντε ώρες έκανε, αλλά πια δεν λειτουργεί, γιατί κανείς δεν θέλει πια να κάτσει πέντε ώρες να κάνει αυτή τη διαδρομή. Οπότε πότε θα κλείσουμε αυτό το κενό της ηλεκτροδότησης. 100 εκατομμύρια τα οποία είναι ψίχουλα σε σχέση με τα δισεκατομμύρια που επενδύουμε σε άλλα πράγματα. Στρασβούργο, Κιέλ, εντάξει, αλλά Φρι, ε, Φράιμπουργκ, με άλλες πόλεις, τι γίνεται. Έχουμε ξεκινήσει επίσης και το One Stop Shop, το σιδηρομικό πακέτο, το οποίο και αυτό εξαφανίστηκε. Γιατί εξαφανίστηκε αυτή η πρωτοβουλία, γιατί λήφθηκε αυτή η απόφαση. Τέλος. Συμφωνώ με το να στηρίξουμε τον προπολογισμό πριν από τις εκλογές. Η κυρία Σαντέρ, ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Να σας πω να σας πω ότι στον προϋπολογισμό να λαμβάνουμε υπόψη μας τη ζήτηση για κονδύλια. Οπότε ρωτάω κατά πόσο μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα χρυσό κανόνα, ένα golden rule, όπου η συγχρηματοδότηση δεν θα έχει οριστικό βάρος και θα επιβαρύνει τα, το δημόσιο χρέο των χωρών μελών. Μετά, για να υποχρεώσουμε με τρόπο λογικό τις χώρες μέλη να τηρήσουν τις ευρωπαϊκές τους δεσμεύσεις. Πώς θα μπορούσαμε, πιστεύετε, να κάνουμε μια αναθεώρηση στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο των υποχρεώσεων για οικοδόμηση ευρωπαϊκών υποδομών. Δηλαδή, να βοηθήσουμε κάπως τις χώρες μέλη, ώστε να κάνουν ακριβώς αυτά που πρέπει. Γιατί ξέρετε ότι τα εθνικά σχέδια δεν έχουν συχνά καμία σχέση ακριβώ με τα ευρωπαϊκά σχέδια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίο ομιλητή, ομιλήτρια, κυρία Ντεμόντα, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλώ ορίσατε, κύριε Επίτροπε. Εγώ θα μιλήσω για τα Βαλκάνια. Συμφωνώ απόλυτα για, με αυτά που είπατε για τη σημασία δηλαδή ολοκλήρωση αυτών των κονδυλίων με τα διαθέσιμα κονδυλία συγχρηματοδότηση με μια νέα λειτουργία, δηλαδή να προωθήσουμε την ολοκλήρωση αυτής της περιοχής. Για τις κοινωνικές κινέζικες επενδύσεις, η Κομισιόν γνωρίζει κατά πόσο είναι αυτά τα κονδύλια τα κινέζικα ε, με ζημιά. Τι γίνεται. Θα θεωρηθούν χαμένα σε κάποια χρόνια. Μιλάμε για υποδομή και μεταφορές, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και Επιτροπή Τουρισμού και ψηφίσαμε ένα ψήφισμα για τη σημασία του τουρισμού και την ε, πρόθεσή του και για την σημασία δημιουργίας ε, μιας γραμμής στον προπολογισμό του τουρισμού. Συμφωνείτε με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δεμόντε Να επανέλθω σε δύο σημαντικά σημεία, λέει η Πρόεδρος, για τον ίδιο προπολογισμό. Ένας προπολογισμός σε σχέση με τις προκλήσεις της Ένωσης θα αρκέσει ή όχι. Αυτό το συζητάτε καθόλου με τις ε, χώρες μέλη. Και μετά, ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι συσχετισμοί σε σχέση με την συμβολή στον προπολογισμό των χωρών. Κάποιοι θέλουν να μην συμβάλλουν παραπάνω. Και τέλος, σε σχέση με τον επαναπροσανατολισμό το δημοσιονομικό, τι γίνεται με τις προκλήσεις για τις οποίες δεν θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια. Ο αντίκτυπο τη κλιματική αλλαγής που θα πρέπει να συνοδεύεται με την κατάλληλη φορολογία, πρώτον και δεύτερον, η ψηφιακή επανάσταση. Η πέμπτη γενιά, το 5G. Αύριο θα είναι παντού αυτή η ψηφιακή επανάσταση. Οπότε, τι γίνεται και εκεί. Σα ευχαριστώ, κύριε Έτιγκερ. Έχετε 8 λεπτά μόνο στη διάθεσή σα για να τηρήσουμε ακριβώ την ώρα την οποία σχολούν οι διερμηνείς. Παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα θέλαμε να υποβάλουμε μια πρόταση για τον προπολισμό, η οποία θα είναι ταυτόχρονα ρεαλιστική αλλά και φιλόδοξη. Αν η Βουλή σας, το σώμα σας. Εδώ, φεύγοντας από εδώ, πάμε στην Επιτροπή Γεωργίας και θα μου πούν δεν θέλω περικοπές, θέλουμε πιο πολλά χρήματα. Πάω σε, άλλο, σε άλλη επιτροπή να μου πούν ότι ας διπλασιάσουμε τα κονδύλια για το 2020 ας πούμε. Όλοι λοιπόν έχουν τις δικές τους απόψεις. Ε, το ίδιο στην εκπαίδευση, πολιτισμό κτλ. Μετά θα πάω στο Συμβούλιο και θα μου πούν κάποιες χώρες μέλη 1% μέγιστο. 1% το πολύ. Οπότε βλέπετε ότι αντιμετωπίζω πια το τετραγωνισμό του κύκλου. Και γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε για πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Κομισιόν είναι λογικό και αναμενόμενο ότι δεν θα μπορέσουμε να εικονοποιήσουμε τους πάντες. Επειδή αυτό αποδεικνύει και εγώ συμφωνώ ότι είναι υπερβολικέ αυτές οι προσδοκίε και κανείς δεν μπορεί να πει ή να ισχυριστεί ότι η πρόταση είναι άδικη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε βέλτιστη χρήση περιορισμένων κονδυλίων που θα έχουμε στη διάθεσή μα. Και ελπίζω εγώ η οροφή να ανέβει κάπως περισσότερο από το 1%. Νομίζω το Κοινοβούλιο προτείνει 1,3%. Και είναι προφανές ότι εσείς στην Επιτροπή μεταφορών, αυτή που ασκείτε την πολιτική των μεταφορών, έχετε προφανώς τα δικά σας και σωστά επιχειρήματα. Ένας προϋπολογισμός, ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν αρκεί για να χρηματοδοτήσει όλες τις υποδομές. Το ΣΕΦ δεν πρέπει να χρησιμοποιεί, ας πούμε, να χρησιμοποιεί τα κονδυλιά του για να χρηματοδοτήσει αυτοκινητοδρόμους ή την ηλεκτροδότηση των σιδηροδρόμων. Αυτό είναι δουλειά του φορέα που λειτουργεί αυτή την υποδομή. Ο οργανισμός ο σιδηροδρομικός της κάθε χώρας ή οποιοδήποτε άλλος. Και οι βουλευτές από την κάθε χώρα ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και τι είναι περισσότερο αποδεκτό. Εμείς εδώ στις Βρυξέλλες είναι αλήθεια ότι είμαστε μακριά καμιά φορά και ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρήσουμε και την αρχή της επικουρικότητας. Το ευρωπαϊκό λοιπόν εξάμεινο μου φαίνεται μια θαυμάσια ιδέα γιατί είναι προφανές ότι αν θέλουμε να ενισχύσουμε μια περιφέρεια ή μια χώρα μέλους, αν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων εργασία εκτός από την δημοσιονομική πολιτική και εκτός από την ποιότητα ας πούμε του εκπαιδευτικού συστήματος θα είναι σημαντικό να ασχοληθούμε και με την υποδομή πέρα από την αγορά εργασίας βέβαια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο όσον αφορά τις συγκεκριμένε συστάσεις αναχώρα θα μπορούσα να πω ότι θα κάνουμε και συστάσεις που θα αφορούν τα δίκτυα μεταφορών ώστε οι αντίστοιχη χώρα μέλος να εγκρίνει μαζί με εμά τις συστάσεις αυτές και μετά να τις συγχρηματοδοτήσει. Εδώ μιλάμε ξεκάθαρα για, την, για τον λειτουργικό επιχειρησιακό προσανατολισμό και νομίζω ότι στη χρηματοδότηση ενός έργου ο κύριος υπεύθυνο, αρμόδιος, είναι η Γενική Διευθύνση MOVE. Έχουμε το εδώ το Γενικό Διευθυντή της. Έχουμε και την κυρία Μπούλτς, η οποία είναι και υπεύθυνη στη στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Για τον έλεγχο του προπολογισμού υπεύθυνο είμαι εδώ. Είμαι εγώ και για το καθαρισμό των προτεραιοτήτων του 2050 θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο το ίδιο το Κοινοβούλιο. Η Ευρωβουλή. Μιλάμε ε, επιχειρησιακά για την Κομισιόν ως Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση. Όμως για τον καθορισμό των, των στρατηγικών προτεραιοτήτων των μακροπρόθεσμων θα πρέπει να αποφασίσουν η Ευρωβουλή και τα Εθνικά Κοινοβούλια οι ευρωβουλευτές και οι εθνικοί βουλευτές. Τώρα, για την χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είμαι αντίθετος, αλλά βλέπω πολλές φορές ότι στο τέλος, όταν κάνουμε τον απολογισμό, πολλές φορές είναι πιο ακριβή αυτή η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα από ότι είναι η δημόσια. Ε, καμιά φορά έχουμε και ψευδεστήσεις, στη Γερμανία μάλιστα. Συνέβη αυτό. Γιατί αν έχουμε μια συνεργασία εξειδικευμένη με μηχανικούς λοιπά, Αν έρχονται όμως να βάλουν χρήματα για να βγάλουν πολύ περισσότερα, τότε απλά και μόνο μιλάμε για αύξηση του κόστους του έργου σε σχέση με χρηματοδότηση του έργου αυτού, το, η οποία θα προερχόταν από το δημόσιο. Η χρηματοδότηση πρέπει να δούμε κατά πόσο έμεσα εμπλέκεται εδώ. Δηλαδή η Βουλγαρία, Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρος, Ιταλία είναι χώρε οι οποίε ε, θίγονται περισσότερο από αυτές τις ε, διαδικασίες. Και η Ισπανία. Και στη χειρότερη περίπτωση θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μάλιστα και για την Πολωνία ή την Ουκρανία. Αλλά θα πρέπει να βρούμε το κατάλληλο μέτρο, την κατάλληλη λύση ελεγγύης. Γιατί αυτό που κάνουν αυτές οι χώρες στη Μεσόγειο από σε κάθε χώρα τεχνικά, οικονομικά δεν μπορεί να το αναλάβει ως έργο, ως βάρος. Γι' αυτό ακριβώς ε, παρεμβαίνουμε εμείς, η Frontex ας πούμε, στον επόμενο ΠΔΠ. Και τέλος, αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία αφορούν στρατιωτική κινητικότητα. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Στην Ευρώπη θέλουμε να μπορούμε να μεταφέρουμε στρατιωτικό υλικό με ταχύτητα από χώρα σε χώρα, ώστε να αντιδράσουμε σε περίπτωση όπου θα χρειαστεί, που ελπίζουμε και ευχόμαστε να με συμβεί ποτέ. Είμαι πεπισμένος ότι αυτός, ας πούμε, που θα περάσει από μια γέφυρα που αντρέχει 60 τόνους, τότε και σε καιρό ειρήνη, φαντάζομαι, αυτή η γέφυρα μπορεί να αντέξει το ίδιο βάρος σε πολιτική κίνηση φορτηγών, αυτοκινήτων, ποδηλάτων κλπ. κλπ. Μιλάμε για υποδομές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε καιρό ειρήνης. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στην στρατιωτική υποδομή, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για πολιτικούς λόγους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τιγκέρ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εξ ονόματος της Επιτροπής μας των Μεταφορών για το χρόνο σας και την τιμή που μας κάνατε να μας δώσετε κάποιες κατευθυντές γραμμές και να έλθει ότι συνεργαζόμαστε καλύτερα και μόνο με αυτή την καλύτερη συνεργασία μεταξύ ημών, Ευρωβουλή, Κομισιών, Εθνικών Κοινοβουλίου θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Και θα πρέπει να σταματήσουμε σε λιγάκι. Πάντως σας χειροκροτούμε. σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Thank you. Alors, mes Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι πήγαμε γρήγορα και να βάλουμε άλλο ένα στοίχημα, θέλετε να ακούσετε. Μια και πήγαμε γρήγορα, μια και έχουμε και δύο-τρία λεπτάκια ακόμα. Να σας πω λοιπόν μόνο να σας πω μόνο ότι βλέπετε ότι το διακύβευμα το δημοσιονομικό του προπολογισμού σας έχει ανάγκη. Θα πρέπει εσείς να κάνετε τα δέοντα στις χώρες σας, όπως και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αποφασισμένη ώστε να υπάρξουν τα απαραίτητα κονδύλια για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών, της λοπής των ευρωπαϊκών δικτύων, δικτύων και των υπολείπων διακυβευμάτων που αφορούν και τις χώρες σας. Υπάρχουν, υπάρχει ένα στόχος να μιλάμε για τις μεταφορές. Δηλαδή, να διευρύνουμε την κινητικότητα, την καθημερινή των πολιτών μας. Αυτό είναι ο στόχος μας και θα πρέπει... Ναι, εντάξει, βεβαίως έχουμε και τα εμπορέματα, το οποίο όμως την επαύριο θα πρέπει να αρχίσουν να μεταφέρονται διαφορετικά. Έχουμε τις καινοτομίε με τα ψηφιακά, τα οποία είναι θαυμάσια εργαλεία για να δημιουργήσουμε καινοτομίε, τις οποίες θα πρέπει να διευρύνουμε και θα πρέπει ο καθένας από εσά από μόνος του να κάνει ανταλλαγές βελτίστων πρακτικών. Οπότε σήμερα εσεί βρίσκεστε στην Ευρωβουλή. Μην διστάσετε να μας προσκαλέσετε στα δικά σας κοινοβούλια την επόμενη φορά, ώστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια από κοινού, ώστε να τα καταφέρουμε μαζί. Ελπίζω πάντως να ήταν καρποφόρο και για εσά το σημερινό απόγευμα και να ξέρετε ότι οι πόρτες της Επιτροπής Μεταφορών του Κοινοβουλίου θα είναι πάντοτε ανοιχτές για σας, τουλάχιστον δύο φορέ το χρόνο, ώστε να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και μην διστάσετε, να μην διστάσουμε μάλλον όλοι ώστε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα θαραλέο και αποφασιστικό προπολογισμό για το θέμα των μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ.